να αναφερθώ σε κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Μίλαν για την Μαυρετανία σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε με την Μαυρετανία για επέκταση κατά ένα έτος της, το πρωτόκολλο της Συμφωνίας Βιώσιμης Αλίας. Αντί για Νοέμβριο 19 έχουμε πάει στο Νοέμβριο του 20. Οπότε αυτά. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι μία από τις δύο συνεδριάσεις που θα γίνει για την κατάσταση των θαλασσών των αλλιευμάτων. Συγκεκριμένα για να σας δώσουμε μία γενική εικόνα στην αρχή της εντολής σύμφωνα με την κοινή αλληλευτική πολιτική για να επιτύχουμε την ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση μέχρι το 2020 και το θέμα είναι βεβαίως ε, τι πρόοδο έχουμε κάνει μετά από 6 χρόνια. Η κυρία Ελίζα Ρόλερ θα μιλήσει πρώτη από την Κομισιόν. Έχετε λοιπόν τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Η παρουσίασή μας έχει δύο μέρη. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια γενική παρουσίαση και μετά η συναδελφός μου η κυρία Κίρχινερ, η αρμόδια για Ατλαντικό και Βαλτική θα αναφερθεί στην κάθε περιοχή χωριστά. Οπότε, πώς ε, έχει η κατάσταση των θάλασσών μας. Είναι, θα έλεγα, ένα έργο εν εξελίξη, διαρκώς. Βγάλαμε μια δήλωση πολιτικής ε, τον Ιούνιο, η Κομισιόν ενέκρινε την ετήσια δήλωσή της που δίνει μια ένδειξη για το πού θεωρούμε ότι πηγαίνει η πολιτική σε σχέση με τους στόχους που έχουν αναφερθεί, μεταξύ των οποίων και υποχρεώσεις εκφόρτωσης, την κατάσταση του στόλου και αυτό το οποίο λέει η δήλωση είναι ότι σε σχέση με τον στόχο του να επιτύχουμε την ε, στη βιώσιμη απόδοση. Η μέση θνησιμότητα έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 1 και έχουμε ορίσει 51 συνολικά επιτρεπτά αλλιεύματα από τα 81 συνολικά. Οπότε όπως σας είπα είναι ένα έργο το οποίο συνεχίζεται και όπως σας είπα η συνάλφος θα σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο βλέπουμε επίσης είναι μια αύξηση στον όγκο της βιομάζας κατά 36% 100 τα τελευταία 15 χρόνια, οπότε βλέπουμε μια βελτίωση. Εάν τώρα δούμε συγκεκριμένα την κάθε περιοχή, στο διάγραμμα βλέπουμε το ποια είναι η αλλιευτική πίεση σε σχέση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Αυτή είναι η γραμμή εκεί στο 1. Η μαύρη γραμμή μας δείχνει την εξέλιξη των δικτών στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Η κόκκινη γραμμή είναι η ελευτική πίεση στον βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό, ενώ το πράσινο μας δείχνει την αλληλευτική πίεση στον βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό εκτός ευρωπαϊκών υδάτων. Η πράσινη γραμμή είναι μη ευρωπαϊκά υδάτα. Η κόκκινη γραμμή είναι ευρωπαϊκά υδάτα. Αν δείτε το απόθεμα τη βιομάζου, που βλέπουμε μία αύξηση κατά 36% βλέπετε ότι οι γραμμές αυξάνουν αργά αλλά σταθερά οπότε η μαύρη γραμμή στη Μεσόγειο και την μαύρη θάλασσα μας δείχνει ελάχιστη έως καθόλου βελτίωση αλλά οι άλλες γραμμές δείχνουν μια σημαντική βελτίωση. Οπότε και πάλι, πώς έχουν τα πράγματα. Η πρόοδος συνεχίζεται Προσπαθούμε να επιτύχουμε τον στόχο αυτό της μέγιστης βιώσιμη απόδοσης. Συνολικός όγκο βιομάζας είναι 36% υψηλότερο και σε σχέση με τον στόλο αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι δυνατότητες του όγκου συνεχίζουν να μειώνονται η χορτικότητα ενώ η οικονομική απόδοση ε, εξακολουθεί να δημιουργεί κέρδη ρεκόρ. Έχουμε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Ε, το οποίο είναι αύξηση κατά 2,7% το έτος. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο βλέπουμε, και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι της ε, πολιτικής ε, αλληλευτικής, είναι η διακυβέρνηση. Βλέπουμε ότι το 2013 είχε μια νέα μορφή διοίκησης, περιφερειακή, με στενή εμπλοκή των ενδιαφερομένων μέσω των συμβουλευτικών συμβουλίων. Τώρα έχουμε τέσσερα πολυετή σχέδια και πολύ ενεργά συμβουλευτικά συμβούλια. Έχουμε λοιπόν τις 73 ε, αυτές ε, συστάσεις από τα υποπτικά συμβούλια και στην συμβουλευτική σκοπιά γινόμαστε ένας μεγάλος παίκτη στην Διεθνή Διακυβερνηστών Οκεανών. Αυτό τη σχετική έκθεση δημοσιεύτηκε και πρόσφατα, οπότε αυτά εν ολίγης, είναι τα βασικά επιτεύγματα και το που βρισκόμαστε σε σχέση με την κατάσταση των θάλασσων. Βεβαίω υπάρχουν κάποιε προκλήσει. Ε, πρώτα απ' όλα, και αυτό το είδατε και στι προηγούμενε διαφάνειε, χρειάζεται περισσότερη πρόοδο για να επιτύχουμε του στόχου για την βιώσιμη απόδοση. Προφανώς ε, αυτή είναι βασική προτεραιότητα και χρειάζεται σαφώς μεγαλύτερη πρόοδος. Το δεύτερο αφορά τις υποχρεώσεις ε, εκφόρτωσης η οποία ετέθη ισχύ το 2019 αλλά όπως ε, έχουμε συζητήσει και με τον κλάδο τους ενδιαφερόμενους χρειάζονται μεγαλύτερες προσπάθειες για την συμμόρφωση αλλά και την συλλογή δεδομένων. Χρειάζεται μια καλύτερη εικόνα για το πώς λειτουργούν αυτές οι υποχρεώσεις και το εάν να βλέπουμε μία μείωση στα ανεπιθύμητα αλλιεύματα και γενικώ αλλαγές στο πώς διαχειριζόμαστε την δραστηριότητα αυτή. Το τρίτο θέμα είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε ε, στους παράγοντες των οικοσυστημάτων με συστήματα διαχείρισης ε, των αλληλευτικών αποθεμάτων, όπως παραδείγματο χάρη με τον Μπακαλιάρο της Ανατολικής ε, Βαλτικής. Έχουμε λοιπόν τις προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων, είτε μιλάμε για τη ρήπανση, είτε για την κλιματική αλλαγή, είτε για την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων ειδών. Πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη εικόνα για το πώς επηρεάζονται και τα αποθέματα και η κατάσταση των θαλασσών και πώς μπορούν να συνεχίσουν να ζουν και οι ψαράδες. Οπότε θα απαιτηθούν περισσότερες προσπάθειες από όλους τους ενδιαφερόμενους για να επιτύχουμε αυτούς τους ε, στόχους κοινή αλληλευτικής πολιτικής και εξυπακούεται ότι ε, προφανώς και το Brexit θα επηρεάσει το πώς προσεγγίζουμε την κατάσταση των θαλασσών. Προτείνω τώρα να επεκταθεί η συνάδελφός μου. Και αν έχουμε την ε, δεύτερη παρουσίαση, παρακαλώ, για να σας τα πει. Ναι, πριν ε, μιλήσετε, να πω στους βουλευτές ότι αν θέλετε να μιλήσετε, μπορείτε να το κάνετε τώρα για να πράγματι ξύπνη Όχι ότι θα σας κοιμήσει η μαγιά. Θέλετε να απαντήσετε, να κάνετε μια ερώτηση τώρα. Τι είναι. Είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Όχι, ε, τότε ας περιμένει. Ναι, ναι, ναι, θα σας δώσω το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας καλέσατε σήμερα στην ε, συνεδρίαση αυτή. Με χαρά μου θα σας παρουσιάσω την κατάσταση κάπως πιο λεπτομερώς στις διάφορες λεκάνες, αλλά πριν ε, ξεκινήσουμε να σας δώσω μια γενική εικόνα για το που βρισκόμαστε συνολικά για τα ευρωπαϊκά έντατα αλλά και για κάποια αποθέματα στα οποία έχουμε αλληλευτικά συμφέροντα, αλλά δεν αποφασίζουμε μόνοι μας. Εδώ πέρα βλέπετε την πρώτη στήλη. Η πρώτη στήλη αντιπροσωπεύει την βιώσιμη και μη βιώσιμη αλληλεία και εδώ πέρα λαμβάνει απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της, δηλαδή η Κομισιόν κάνει μια πρόταση και αποφασίζει το Συμβούλιο των Υπουργών. Βλέπετε λοιπόν ότι ο αριθμός των εκφορτώσεων είναι αρκετά ψηλός ε, για αποβιώσιμα αποθέματα, μιλάμε για ένα 98% πιθανότατα ε, που προέρχονται από αποθέματα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και μετά τα μπλε είναι αυτό το οποίο είναι σε κοινή διαχείριση με την Νορβηγία και το άλλο αφορά τις παράκτιες χώρες. Έρχομαι λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Εδώ πέρα βλέπετε τον ε, αριθμό αποθεμάτων ε, που αλλιεύονται βιώσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 50 από τα 57. Τι σημαίνει αυτό. Αυτός είναι ο αριθμός μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ε, που λαμβάνουμε σύμφωνα με το ISIS, δηλαδή το Διεθνές Συμβούλιο για την Διαχείριση των Θαλασσών ε, θεωρεί ότι διαχειριζόμαστε άριστα 50 από τα 57 αποθέματα. Από αυτά τα 57 έχουμε, όπως είπα, πετύχει μέγιστη βιωσιμή απόδοση για τα 50. Ένα αρκετά καλό επίτευγμα, θεωρώ, και τώρα περνάμε στις διάφορες λεκάνες. Ξεκινάω με την Βαλτική, μετά θα δούμε την Βόρεια Θάλασσα και μετά τον Ατλαντικό. Στην Βαλτική το 2019 Έχουμε ε, επιστημονικές συμβουλές για 8 το θέματα. Από αυτά τα 8, τα 7 ε, όσον αφορά τις ε, ποσοστώσεις συμμορφωνόμαστε με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ποιες είναι λοιπόν οι προβληματικές υποθέσεις εκεί πέρα στη Βαλτική. Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε κάποια προβλήματα το ένα απόθεμα το οποίο δεν πετυχαίνει τον στόχο είναι η ρέγγα της Δυτικής ε, Βαλτικής ε, σημαντικό ψάρι και ε, δυστυχώς υπάρχει μια τυχή περίπτωση γιατί δεν υπήρχε ένα πρόβλημα μέχρι το 2018. Το 2018 μας είπαν οι επιστήμονες ότι τα ψάρια δεν ήταν τόσα όσα νομίζαμε και μας είπαν ότι είναι μεγάλη αλληλευτική πίεση οπότε η Κομισιόν έπρεπε να κάνει μια πολύ δύσκολη πρόταση για να μειωθεί η αλία κατά 65%. Έγινε αυτή η πρόταση σύμφωνα με το πολιετές σχέδιο για την Βαλτική ε, το οποίο συντάξατε εσείς μαζί με το Συμβούλιο των Υπουργών και μετά το αποτέλεσμα στο Συμβούλιο ήταν μια περικοπή της ποσόστοσης στο μισό. Οπότε απέκλεινε κάπως ε, το Συμβούλιο από την πρότασή του Κοινοβουλίου. Μετά έχουμε και άλλα ψάρια που είναι επίση καψοβληματικά. προβληματικά. Όπω είπα, η ρέγκα τη Δυτική Βαλτική είναι το μόνο ψάρι το οποίο δεν έχει επιτύχει τον στόχο για το 2019. Μετά πηγαίνουμε στον ε, μπακαλιάρο τη δυτική ε, Βαλτικής, ε, σημαντικό στην Βαλτική και ενώ αυτή τη στιγμή αλλιεύεται σύμφωνα με τον στόχο δεν τον έχουμε επιτύχει ακόμα. Είναι ένα ψάρι που υφίσταται μεγάλε διακυμάνσει τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν πετύχει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση γιατί ε, μεταβάλλονται συνεχώ οι επιστημονικέ συμβουλέ και η βιομάζα. Οπότε, αν ρωτήσετε τι πρέπει να κάνει η Κομισιόν και το Συμβούλιο, οπωσδήποτε αυτό το ψάρι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο έτσι ώστε να μειωθεί η αληφτική πίεση και να έχουμε παραδείγματος χάρη κάποιες ε, ποσοστώσεις επί του γόνου και άλλα τέτοια μέτρα. Και τέλος ε, για τον μπακαλιά της Ανατολικής Βαλτικής, αυτό είναι γνωστό ότι είναι μια μεγάλη ανησυχία στην Κομισιόν και για το Κοινοβούλιο και για τα κράτη-μέλη γιατί ε, δυστυχώς ε, αναγκαστήκαμε να λάβουμε καταπήγοντα μέτρα και να απαγορευτεί τελείως η αλία. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν είναι το εξή άλλη μια τυχή περίπτωση. Βλέπετε μια φωτογραφία ενός τέτοιου ψαριού. Ε, δεν μοιάζει με μπακαλιάρο. Είναι ε, μια εικόνα ενός ε, ψαριού που μοιάζει με μικρό πελαγικό ψάρι. Οπωσδήποτε η υπεραλίευση βοήθησε, είχαμε ορίσει πολύ υψηλές ποσοστώσεις, πρέπει να το παραδεχτούμε, και αρνητικές περιβαλλοντικές εξελίξεις, η θερμοκρασία της θάλασσας, η αλμυρότητα του νερού πολύ χαμηλή, έχουμε ευτροφισμό από τα ζωτούχα, λιπάσματα και επίσης παράσιτα από τις φώκες. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε τα επόμενα χρόνια. Ε, περνάμε λοιπόν στην Βόρεια Θάλασσα και εδώ πέρα βλέπετε τα αλλιεύματα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τα αλλιεύματα στα οποία μπορούμε εμείς να κάνουμε πρόταση ως Κομισιόν και αποφασίζει το Συμβούλιο. Έχουμε μια αρκετά καλή εικόνα εδώ πέρα γιατί και τα 8 είναι εντός ε, των ορίων ε, και αυτά τα όρισε πέρσι το Συμβούλιο σε ένα επίπεδο που σέβεται την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Τώρα ερχόμαστε άρα στον Ατλαντικό και εδώ πέρα η εικόνα είναι κάπως διαφορετική. Βλέπετε πως είχαμε Παρακολουθούμε 41 ήδη, 35 επέτυχαν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Τώρα, ποια είναι τα προβληματικά ήδη Είναι κυρίως ε, στην Κελτική θάλασσα, δηλαδή δυτικά της ε, Σκοτίας. Οι δυσκολίες ε, που έχουμε εδώ είναι ότι δεν έχουμε ακόμα πετύχει την επιλεκτική αλληλεία. Το πρώτο, το ψάρι, ο βακαλάος της Κελτικής θάλασσας εντάσσεται στο σχέδιο των δυτικών υδάτων που μόλις ετέθην ισχύει την Άνοιξη, πολύ σημαντικό αλίευμα και εδώ πέρα ε, η ΆΙΣΙΣ μας λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε τελείως ε, την αλληλεία του χρόνου και να επιτύχουμε βεβαίω μέχρι το 2020 το μέγιστο ε, βιώσιμο αλίευμα. Και το άλλο είναι δύο είδη ενός ψαριού που λέγεται προσφυγάκι στην δυτικά της Σκωτίας και στην Ιρλανδική θάλασσα και αυτά δεν επιτυχάνουν το στόχο ε, είναι αυτά τα οποία λέμε παρεμπίπτοντα αλλιεύματα. Δηλαδή δεν είναι αυτά τα ψάρια τα οποία ψαρεύουν. Ε, οι ψαράδες δεν κυνηγάνε αυτά τα ψάρια, αλλά τα πιάνουν παρεπιπτόντος. Ε, οπότε όταν απλώνουν τα δίχτυα, τα μαζεύουν, μπορεί να θέλουν κάποιο άλλο ψάρι, αλλά πάντα θα έχουν ε, και κάποια άλλα παρεμπιπτοντά αλλιεύματα. Αυτό είναι λοιπόν το δύσκολο. Τι κάνουμε εδώ. Και εδώ πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα, να βρούμε τρόπους να ψαρεύουμε πιο επιλεκτικά, να μειωθεί η αλλιευτική πίεση, εκεί όπου υπάρχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, παραδείγματος χάρη αλλιευμάτων, που πιέζονται. Μετά, τα τελευταία δύο, επίσης ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, δύο είδη ρέγκας, δύο αποθέματα μάλλον Το ένα είναι ε, στα νότια δυτικά της ε, Σκοτίας και εδώ πέρα ο αρμόδιος φορέας μας λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε τελείως την αλληλεία και αυτό το οποίο κάναμε ως κομισιόν είναι να ρωτήσουμε τους επιστήμονες είναι καλύτερο να σταματήσει τελείως η αλληλεία ή να μπει η λεγόμενη επιστημονική ποσόστοση μια μικρή ποσόστοση δηλαδή που χρησιμοποιούν ε, τα επιστημονικά Ινστιτούτα σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. βλώνουν ένα λευτικό σκάφο, ψαρεύουν και συλλέγουν δεδομένα. Ο ε, επιστημονικό οργανισμό μα είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χαθούν αυτά τα δεδομένα. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνο αν σταματήσει τελείω η ελεία, να μην συλλέγονται δεδομένα. Έρχομαι τώρα στο τέλος της παρουσίασης αυτής. Και βεβαίω ευχαρίστω να απαντήσω σε ερωτήσει σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Έλλης, μας ε, παρουσιάσατε 59 από 81 τάξ που είναι ε, σύμφωνα με το στόχο του MSY, αλλά από ό,τι μας είπατε δεν βγαίνουν τα νούμερα. Πώς τα συνδυάζετε την ευρύτερη εικόνα με την τοπική εικόνα. Κοιτάξτε, τα νούμερα που βλέπετε εδώ, 59 από τα 81. Εάν δείτε την πρώτη στήλη, αυτό ε, αντιπροσωπεύει μόνο τα αλλιεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε 50. Και μετά η ισορροπία δυστυχώς πάει προς τα αρνητική πλευρά με τις άδειλες δύο στήλες που βλέπετε εκεί. Έχουμε στόκ όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποφασίσει μόνη της, αλλά εξαρτάται από την καλή θέληση τρίτων χωρών ώστε να ορίσουν τα όρια σε ε, βιώσιμα επίπεδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πριν δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους, λέτε ας πούμε ότι ε, ε, με την Νορβηγία. Η Νορβηγία θέλει να υποτίθεται να ψαρεύει βιώσιμα, ενώ όταν μιλάμε για τα στόκ οι σχέσεις μας δεν είναι καλές, στις διαπραγματεύσεις δηλαδή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φοβούμαι πω είναι λίγο πιο περίπλοκο το θέμα. Η δυσκολία που έχουμε με την Νορβηγία είναι ότι δεν έχουμε την ίδια νομική βάση για την κοινή αλληλευτική πολιτική και ούτε προσεγγίζουμε τον ίδιο τρόπο τη στρατηγική διαχείριση. Η δυσκολία στη συζήτηση είναι ότι βεβαίω καταρχά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα συμβούλιο που στηρίζει πλήρω ε, την πρόταση τη Κομισιόν και όπω υπόθηκε μπορεί να συμβεί σε άλλε περιπτώσει να μην ισχύει κάτι τέτοιο και Πλέον, όταν διαπραγματευόμαστε με την Νορβηγία για αυτό το πλαίσιο, δεν έχουμε πάντοτε την ίδια ε, γνώμη ε, περί στόχου για το συγκεκριμένο απόθεμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτός ο πίνακας που βλέπετε και είναι μια από τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε, ε, ειδικά εκεί όπου έχουμε άμεση συσχέτιση με το στόκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μερίδιο της Ένωσης. Και τέλος, δυτικά ύδατα. Θα μας παρουσιάστηκε για τα δυτικά ύδατα κάτι. Sorry, on the western waters. Για τα δυτικά ύδατα μπορούμε να πάμε πίσω στις διαφάνειες, οπότε βλέπετε εδώ. Εδώ έχουμε τα δυτικά ύδατα. Έχουμε δηλαδή 35 βιώσιμα αποθέματα από τα 41. Θεωρητικώς Έχουμε τη συμβουλή του ISS για, τις, ε, για το MSY, την μέγιστη βιώσιμη απόδοση και εκεί μπορούμε να επιτύχουμε μέχρι εκεί. Προσπάθησα να σα εξηγήσω γιατί το επιτύχαμε, ίσως να μην ήμουν σαφής, να πάω πίσω δηλαδή, να σας εξηγήσω. 35 από 41 στόκ. Αυτά είναι τα 6 στόκ από θέματα για τα οποία δεν έχουμε καταφέρει τους στόχους. MSY. Να αρχίσω από κάτω για τα δύο αποθέματα θέματα ε, Εδώ λέει καθόλου αλία. Ε, πρέπει να σταματήσουμε την αλίευση αυτών των στόκ. Αυτό που κάναμε ήταν, ε, τους ε, καλέσαμε και τους είπαμε, τι κάνουμε, σταματάμε τελείως την αλληλεία ή να ρωτήσουμε τους επιστήμονες αν θα ήταν καλό να έχουμε ένα επιστημονικό τάκ δηλαδή ένα τάκ για επιστημονική αλληλεία. Και επίσης τους ρωτήσαμε ποιο είναι επίπεδο αυτού του επιστημονικού τάκ. Πριν από λίγα χρόνια μας είπαν, εάν θέλετε να κάνετε επιστημονική αλληλεία και θεωρείτε πως είναι σημαντικό και εμείς είπαμε ναι, θεωρούμε πως είναι σημαντικό γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε τα υπόλοιπα στοιχεία και αυτό είναι πάντοτε ένας κίνδυνος Αν σταματήσεις τελείως την αλληλεία, χάνεις τα στοιχεία. Αυτό μας, το, μας είπαν ότι είναι μια χρονική σειρά. Δηλαδή, αρχίζουμε να συλλέγουμε στοιχεία το 1985 και το 1993, 8 χρόνια αργότερα, ξέρεις τι συμβαίνει με το απόθεμα. Και εάν υπάρχει ρήξη σε αυτή τη χρονική σειρά, οι επιστήμονες λένε κάποιες φορές ότι δεν μπορούν να είναι βέβαιοι. Και άρα, από εκεί που υποτίθεται ότι είμαστε ε, στο ανώτερο σημείο, δηλαδή κοντά στο στόχο, ξανακατεβαίνουμε πάλι στην αρχή. Έχουμε λοιπόν επιστημονικές ποσοστώσεις για αυτά τα δύο στόκ. Γι' αυτό και δεν αναφέρουμε αυτά τα δύο αλλιεύματα, γιατί η συμβουλή του ISIS ήταν σαφής ότι δηλαδή δεν πρέπει να σταματήσει τελείως η αλλιεύση. Για το 3 και το 2, εδώ είναι παραλλιεύματα αυτά τα αποθέματα. Ε, αν μιλήσουμε για μια υποθετική κατάσταση. Δηλαδή, τι θα συνέβαινε αν είχαμε μηδενικέ ποσοστώσεις για το... για το προσφυγάκι στα δυτικά της Σκωτίας θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί. Δεν θα πρέπει καθόλου να λιεύονται αυτά τα τρία είδη. Δηλαδή το προσφυγάκι δυτικά της Σκωτίας, το προσφυγάκι στην ε, θάλασσα της Ιρλανδίας και ο γάδος στη, δυτική, ε, στη δυτικά της Σκοτίας. Όμως, όταν κανείς στοχεύει σε υγιείς, ε, υγιή αποθέματα που είναι πιστοποιημένα, που είναι σε βιώσιμα επίπεδα, δεν μπορείς να αποφύγεις τα παραλιεύματα σε προσφυγάκι ή γάδο. Δηλαδή, αν είχαμε αυτές τις ποσοστώσεις στο μηδέν, τότε θα έπρεπε να σταματήσουν και όλα η αλίευση των άλλων βιώσιμων ε, ε, αποθεμάτων. Δηλαδή, να μην υπάρχει καθόλου ε, δυνατότητα λήψης ούτε για τον Ισπανικό στόλο, ούτε για τον Πορτογαλικό στόλο. Ε, θα έπρεπε να σταματήσει τελείως η αλληλεία όλων των ειδών που αλλιεύονται σε αυτά τα ύδατα. Άρα πρέπει να, κάνουμε, να, βρούμε μια συμβιβαστική λύση εδώ. Και αν δούμε το νέο πολιετές ε, σχέδιο που συμφωνήθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εκεί υπάρχει ένα άρθρο που ορίζει ότι οι ε, αλλιευτικές ευκαιρίε θα πρέπει να ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Δηλαδή, εάν είναι μηδέν για το πρώτο ψάρι, ας πούμε, σε αυτόν εδώ τον κατάλογο, θα έπρεπε να σταματήσει η αλληλεία για χιλιάδες αλλιευτικά σκάφη στο Βόρειο Ατλαντικό. Δηλαδή θα ήταν ε, στην ουσία σαν να πηγαίνουμε αντίθετα με το πολιετές ε, σχέδιο. Αυτά είναι τα αποθέματα λοιπόν όπου δεν έχουμε ακόμα επιτύχει την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, το, το MSY. Για το μέλλον πρέπει να ε, επιτείνουμε τις προσπάθειές μας, να βρούμε πώς μπορούμε να γίνουμε πιο επιλεκτικοί και πιο βιώσιμοι. Ακόμα και αν δεν είναι δυνατόν να έχουμε απόλυτα καθαρή αλία, είναι δυνατόν αυτά τα παραλιεύματα να μειωθούν στο απόλυτο ελάχιστο, ώστε να μπορούν να αλλιεύονται τα υπόλοιπα αποθέματα. Αυτά ήθελα να σας πω και φυσικά αν έχετε και άλλες ερωτήσεις ευχαρίστω να σας απαντήσω. Μπορείτε να μας δώσετε μια περίληψη, μια γενική εικόνα για την πρόοδο που έχει γίνει ή δεν έχει γίνει από τότε που ξεκίνησε η νέα αλληλευτική πολιτική το 2013. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί εν γέννη είναι όταν ξεκινήσαμε να μετράμε πόσα βιώσιμα αλλιεύματα είχαμε. Αυτό ξεκίνησε το 2009 και τότε καταγράψαμε 5 αποθέματα. Από πέντε έχουμε φτάσει στα 59 το 2019. Είναι αρκετά καλό επίτευγμα. Αλλά και πάλι Ξέρω που μας, μας αρέσουν να δημοσιεύουμε αυτά μας τα επιτεύγματα, αλλά να γνωρίζουμε πως δεν τα έχουμε καταφέρει απόλυτα ακόμα, ούτε μπορούμε να αναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Γι' αυτό Ακόμα και για τα υγιή αυτά αποθέματα, η κατάσταση μπορεί να ανάξει του χρόνου ή του παραχρόνου. Ε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τη φύση. Ένα χρόνο μπορεί να έχουμε πολλά, ε, πολλά, ε, πολλούς νεογνούς και τα αποθέματα για δύο-τρία χρόνια να είναι καλά, αλλά για τρία-τέσσερα χρόνια μετά να μην έχουμε τις ίδιες γεννήσεις. Οπότε να ξαναμειωθεί το στόκ. Πρέπει να ακολουθήσουμε, να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτό το μονοπάτι MSY μαζί με το πολιετές πλάνο για αυτά τα βόρεια ύδατα, με τη λήψη αποφάσεων πολλές φορές μπορεί να είναι σκληρές αποφάσεις. Ας πούμε για του χρόνου η Κομισιόν έχει υποβάλει πρόταση λίγες μέρες πριν μάλιστα για τις ποσοστώσεις της Βαλτικής θάλασσας και εκεί έπρεπε να προτείνουμε τη μείωση πάλι ε, κατά τα 3 τέταρτα 71% την αλίευση της ρέγας της Δυτικής Βαλτικής γιατί η Άισες είπε ότι δεν ήταν δυνατό να συνεχίζεται η αλίευση αυτού του είδους ε, ε, εφόσον θέλουμε το αποθεματικό να αναγεννηθεί και να αναπληρωθεί για την Παπαλίνα έπρεπε επίσης ε, να προτείνουμε περικοπή ε, των ε, δυνατοτήτων αλίευσης. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντάλεν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις δύο κυρίες. Υπάρχουν δύο ερωτήματα που είχα. Η κυρία Ρόλερ αναφέρθηκε κάπως ε, στην υποχρέωση ε, εκφόρτωσης. Ε, βεβαίως το θέμα είναι ακριβώς τα ίδια εκείνα τα οποία κινδυνεύουν με πνιγμό, ασφυξία μάλλον, και θα πρέπει ακριβώς ε, να υπάρξει ένα σταμάτημα της αλίας τους. Ε, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας διαγραφίσετε πώς έχουν, πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες ε, στενοποί ή θεωρείτε ότι η κατάσταση είναι λιγότερο δραματική από ό,τι είχαμε εκτιμήσει. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όταν μιλάμε για συγκεκριμένα είδη, θα ήθελα να δούμε την ε, κατάσταση της γλώσσας ε, στη Βόρεια Θάλασσα. Βλέπετε ότι αφενός η οργάνωση ISIS λέει ότι η κατάσταση είναι αρκετά καλή με την γλώσσα. Από την άλλη βλέπουμε ότι τα αποθέματα της ε, γλώσσας σχεδόν έχουν εξαντληθεί. Αν δούμε στην Ολλανδία έχουμε εξαντλήσει σχεδόν τη μισή ετήσια ποσόστοση και βλέπουμε ότι σε όλους τους αριθμούς ε, η γλώσσα εξαφανίζεται. Θα ανέμενε κανείς ότι με την ε, νέα πρόταση ποσόστοσης ε, δεν θα είχαμε κάποια μείωση της γλώσσας, αλλά μιλάμε πάλι για μείωση κατά 8% στην ποσόστοση της ε, γλώσσας, κάτι το οποίο δεν ε, ταιριάζει με την ε, πρακτική. Πράγματι μπορεί να σχετίζεται αυτό με τη θερμοκρασία του νερού, αλλά από φαίνεται οι επιστήμονες μας λένε ότι ναι, πάνε καλά τα πράγματα με την γλώσσα, αλλά θέλουμε να διατηρηθεί. Οι απ' την άλλη οι ψαράδες λένε δεν ψαρεύουμε αρκετά και δεν εξαντλούμε την ποσόστοση. Υπάρχει λοιπόν μια τριβή αφενός επιστημόνων και αφετέρου ψαράδων και η σχέση μεταξύ των δύο είναι κάπως τεταμένη. Οπότε αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις. Το ένα υποχρέωση εκφόρτωση και το άλλο γλώσσα. Ευχαριστώ. Okay, we'll take two or three together. Mrs. Mummery. Thank you, Chairman. We have heard a lot of talk about... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά για συγκεκριμένες περιοχές. Παρόλα αυτά, είναι ένα σημαντικό κομμάτι που έχουμε παραβλέψει κατά πόσο φαίνεται το Ηνωμένο Βασίλειο θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας τα δικά μας αποθέματα θα μπορούσατε να μου πείτε αν η Επιτροπή αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη διαπραγματεύονται όλα αυτά τα μέτρα διατήρησης και κάποιες πιθανές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο σαν εξάρτητο κράτος. Επίσης, μπορείτε να μου πείτε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να προχωρήσει πάνω στο θέμα αυτό με μια καινούρια ανεξάρτητη κυβέρνηση, ακολουθώντας ένα no-deal Brexit μετά την 31η Οκτωβρίου. Να επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι όλη η δουλειά σας θα είναι ξεπερασμένη. Έχετε τα ίδια δεδομένα με το Ηνωμένο Βασίλειο ξεχωριστά ως ανεξάρτητο κράτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλαντ. Άκουσα σήμερα το πρωί, είπατε ότι επισκεφτήκατε κάποιους αλληλευτικούς οργανισμούς και θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ για τον βακαλάο στη Βόρεια Θάλασσα. Ακούμε πολλά από τους διάφορους οργανισμούς που λένε ότι δεν υπάρχει ένα και μόνο σωστό μέγεθος αποθέματος και αυτό είναι μια τεράστια συζήτηση σε ό,τι αφορά τον βακαλάο. Υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα για τα αποθέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε και στην πραγματικότητα. Δεν ξέρουμε επακριβώς τι συμβαίνει. Χάρηκα σήμερα που συζητήσαμε για τα, παράθ, για τα παράσετα, που συζητήσαμε και για την αλληλευτική πίεση και για την χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα. Αυτό που θα ήθελα να ακούσω όμως σήμερα και σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε από τον Άισις, καθότι ακούσαμε ότι μπορεί και να μην είναι απολύτως ακριβή, θα ήταν δυνατόν στο μέλλον να έχουμε κάποια άλλα συστήματα, να έχουμε ένα διαφορετικό μοντέλο να, ή να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε αυτό που έχουμε τώρα, διαφορετικά συστήματα, για να έχουμε μια διαφορετική εξέταση των στόκ, των αποθεμάτων. Το δεύτερο σημείο τώρα που θέλω να θίξω, θέλω να μιλήσω πιο συγκεκριμένα ε, για τα σειρώμενα σκάφη που αλλιεύουν ε, βακαλάους. Και θα ήθελα, και για τα δίχτυα πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο αυτό το ζήτημα προκειμένου να μην καταλήξουμε σε μια καταστροφή. Θα ήθελα η Επιτροπή, όπως είπε και ο Φιλανδός υπουργό, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν φεύγει ακόμα και μπορεί και να μην φύγει. Αν δεν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο θα δούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Σήμερα ακούσαμε ότι δεν έχουν φύγει προς το παρόν. Και θέλω η Επιτροπή αυτή να το λάβει υπόψη της ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει φύγει. Μπορεί και να μην φύγει, επομένως και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας από εδώ και στο εξή. Άλλη μία ερώτηση και θα ζητήσω στη συνέχεια από την Επιτροπή να απαντήσει. Απλώς να πω ότι ο κύριος Άλλαντ μίλησε για διαφορετικά μοντέλα. Νωρίτερα είπα ότι ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε προσκεκλημένους εδώ και το ISIS να μας εξηγήσουν κάποια πράγματα παραπάνω κατά πόσο μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις εκτιμήσεις τους κτλ. Επομένως, αν τα ερωτήματά σας έχουν καλυφθεί ήδη από αυτή την παρουσίαση. Άκουσα με πολύ προσοχή ε, σε εκπροσώπους της Κομισιόν και ε, μάλιστα διάβασα και το ανακοινωθέν και σας ευχαριστώ και αυτό και μάλιστα ε, ε, ίσως θα έπρεπε να δοθεί και δημόσια διαβούλευση αυτό το θέμα για τις δυνατότητες για το 2020 πριν οριστούν τα τάκα και οι ποσοστώσεις. Αυτή η διαβούλευση ε, της ανακοίνωσης αυτής ε, είναι πολύ σημαντική για να δούμε και τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο αυτών των προτάσεων. Θα ήθελα να διαπιστώσουμε ότι μετά από πολλές προσπάθειες και συμβιβασμούς από πλευράς ε, του αλληλευτικού τομέα καταφέραμε κατάφεραν έναν, ε, σε μια σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή τα νούμερα που είδαμε, τα ποσοστά σε σχέση με τα ΤΑΚ, βλέπουμε πως έχουν φτάσει τα πολλά αποθέματα σε βιώσιμο επίπεδο και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο γιατί ε, μόλις πριν 10 χρόνια τα νούμερα των αποθεμάτων και των ΤΑΚ ήταν ε, ε, πολύ μικρότερα. Ήταν πέντε μόνο τα αποθέματα ε, τα ληφτικά, ενώ τώρα είναι 59. Πολύ μεγάλα και θεματικά. σπουδαία ε, αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, να μην επαναπαυθούμε, να μην κάνουμε άλλες προσπάθειες. Υπάρχουν κάποια στόκο που είναι σε κακή κατάσταση. Ε, το θέμα του, ε, ανατολικής, του, του γάδου της Ανατολικής Βαλτικής θάλασσας, ε, αλλά γενικά είναι θετική εικόνα. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν θα οριστούν οι ποσοστώσει το Δεκέμβριο. Εγώ μάλιστα σήμερα το πρωί το είπα και στον Υπουργό των Φιλανδό της Προεδρίας ότι θα πρέπει ε, η βελτίωση των στόκ να έχει αντίκτυπο και στις ποσοστώσεις που θα οριστούν. Αυτό κατέστη δυνατόν και ε, ε, λόγω της μείωσης των αλευτικών σκαφών. 22.000 σκάφη λιγότερα έχουμε και αυτό παρατηρείται. Ε, και τα αποθέματα που ήταν σε πολύ κακή κατάσταση έχουν ε, δει μεγάλη βελτίωση. Στην Μεσόγειο είναι χειρότερη η κατάσταση, αλλά πιστεύω πως το θέμα της κατάστασης της αλληλείας στην Μεσόγειο δεν είναι μόνο θέμα υπεραλήψης, υπάρχει και το θέμα ε, το περιβαλλοντικό, κλιματική αλλαγή κτλ. Έλεγα λοιπόν ότι για τον ορισμό των ε, ποσοστώσεων αυτά τα ελπιδοφόρα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά και το γεγονός που προηγουμένως ανέφερε η εκπρόσωπος ε, της Κομισιόν της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αποφεύγουμε να δημιουργούνται τέτοιες ε, καταστάσεις με τα παραλιεύματα και την υποχρέωση εκφόρτωσης. Δηλαδή, όχι επειδή έχουν πολλά παραλιεύματα τα σκάφη να πρέπει να γυρνάνε στο λιμάνι άπρακτα, ε, θα πρέπει κάπως να δούμε αυτό το μέτρο. Είναι μια πραγματική επανάσταση, η υποχρέωση εκφόρτωσης, η, απαγόρευση της ε, ε, ρήψη στη θάλασσα είναι μεγάλη επανάσταση. Τώρα, δεν θα ήθελα, όπως πιστεύω και οι περισσότεροι από εμά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι τα στόκ τα οποία μοιραζόνται οι Ευρωπαίοι τη υπηρετικής Ευρώπης με τους Βρετανούς. Έχουμε αυτό το Brexit, όμως θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να διαχειριστούμε από κοινού τα αποθεματικά. Η Κομισιόν θα πρέπει αυτό να το γνωρίζει ότι σε περίπτωση που γίνει το Brexit, που επαναλαμβάνω εγώ δεν το επιθυμώ, θα πρέπει όσο γίνεται νωρίτερα να φτάσουμε σε συμφωνίες που θα μας επιτρέπουν αμοιβαία πρόσβαση στα ύδατα και στους πόρους. Το Brexit δεν μπορεί να είναι ένα σκληρό διαζύγιο, αντίθετα θα πρέπει να είναι μια νέα μορφή συνεργασίας όπου η Αλία θα πρέπει να έχει εξέχοντα ε, ρόλο. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε. Η κυρία Κίρσνερ, η κυρία Ρόλερ, θέλετε να απαντήσετε σε αυτό το πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ναι, ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με το ερώτημα του κυρίου Φαντάλεν για τη Βόρεια Φάλαση και την αλία χωματίδας εκεί. Σύμφωνα με τη συμβολή του ΆΙΣΕΣ, που είναι η καλύτερη συμβολή που έχουμε στα χέρια μας, θα πρέπει σιγά σιγά να μειώσουμε την αλία της χωματίδας, μείον 8%. Ρωτήσατε πώς είναι αυτό δυνατό. Αν οι ψαράδες μας μας λένε ότι δεν ε, φτάνουμε καν το ποσοστό, δεν φτάνουμε καν το 50% του ποσοστού που μας αναλογεί. Η χωματίδα είναι ένα αρκετά ευαίσθητο είδος. Οι, οι ψαράδες δεν θέλουν να ψαρεύουν αυτό το ψάρι, προτιμούν να ψαρεύουν ε, αντιθέτω γλώσσα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να ψαρέψουν μόνο τη γλώσσα χωρίς να ψαρεύουν παρεμπιπτόντως και χωματίδα. Άρα θα πρέπει να μειωθεί κατά 8% η ποσόστοση της χωματίδας. Και αυτό που μπορώ να σας πω από την πλευρά μου είναι ότι η μοναδική καλύτερη συμβουλή που έχουμε και αυτή είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Και τουλάχιστον αυτό είναι αυτό το οποίο θα προτείνει η Κομισιόν, εμείς ακολουθούμε τις συμβουλές του ISIS για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση σε ό,τι αφορά το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι που το ISIS προτείνει να μειωθεί η αλία, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί, διαφορετικοί λόγοι, αλλά το ISIS πάντοτε μα δίνει τι συμβουλέ του με βάση τα τελευταία δεδομένα. Αν λοιπόν μα λένε το απόθεμα φέτο είναι λίγο μικρότερο από ό,τι ήταν πέρσι, τότε αυτό έχει αντίκτυπο στη συμβουλή που προτείνουμε και εμεί με τη σειρά μα. Εάν μα πούνε ότι η αλευτική πίεση είναι μεγάλη, πάλι θα μα πούν να ψαρέψουμε λίγο λιγότερο. Όλε αυτέ οι πληροφορίε βρίσκονται στη συμβουλή που μα δίνει το ISIS και αυτό είναι αυτό το οποίο ακολουθούμε εμεί και καταλήγουμε στο μείον 8%. Να απαντήσω τώρα απευθείας στην ερώτηση του κυρίου Άλλα. Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε διαφορετικά μοντέλα όταν υπολογίζουμε τα αποθέματα. Ε, πραγματικά με ενδιαφέρει η ερώτησή σας, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που θίξατε. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε κάποια αποθέματα σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, σύμφωνα με το νέο σχέδιο των δυτικών υδάτων και οι ποσοστώσει για τα λιεύματα αυτά είναι πολύ ψηλές. Αλλά μέχρι στιγμής το ISIS μας δίνει προληπτικές συμβουλές. Και εμείς θα πρέπει να διαχειριστούμε τα προϊόντα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε συνεργασία με το ISIS. Επομένως πρέπει να μιλήσουμε με τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη που έχουν την μεγαλύτερη παρουσία στην αλληλεία των ψαριών αυτών ε, να μας πούν κατά πόσο έχουν το απαιτούμενο προσωπικό, κατά πόσο έχουν τους οικονομικούς πόρους για να ερευνήσουν κατά πόσο τα αποθέματα αυτά που, για, για, τα οποία το ISIS δεν μπορεί ακόμη να μας δώσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, μια συμβουλή μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Ελπίζω αυτό να απαντάει το, στο ερώτημά σας. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Ελίζα. Σε σχέση λοιπόν με την ερώτηση του κυρίου Βανταλέν για την υποχρέωση εκφόρτωσης το ερώτημα των αλευμάτων υποπίεση είναι κάτι το οποίο συνδέεται στενά από την αρχή με την υποχρέωση εκφόρτωσης. Βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις με αρχές ελέγχου, με μπλεκόμενα μέρη, ούτω ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ομαλή εφαρμογή του μέτρου αυτού και πιο συγκεκριμένα προσπαθούμε να ασχοληθούμε με αυτά τα είδη υποπίεση. Υπάρχει ένα choke tool, ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να μελετούμε πιο συγκεκριμένα στην Βόρεια Θάλασσα Πέρσι είχαμε και κάποιες ποσοστώσεις που αφορούν στην παρεπιπτόντος αλληλεία, στα, στα, στα, είδη που παρεπι, στα είδη που αλλιεύονται, με συγχωρείτε, παρεπιπτόντω, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοιου τύπου α, περιπτώσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε επίσημη αναφορά, υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες, δεν έχουμε μια επίσημη α, αναφορά, αλλιευμάτων που να έχουν, ε, ειδών που να έχει πάυσει η αλία τους λόγω τέτοιου τύπου πίεσης. Όπως σας είπα και πριν, υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο προ, προόδου σε ό,τι αφορά την υποχρέωση εκφόρτωσης, κυρίως σε ό,τι αφορά την καταγραφή και την απόρριψη. Και δεύτερον, υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα συμμόρφωσης, ε, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού με τις αρχές ελέγχου σε σχέση με τον κύριο Μιγιαν Μόντορε και την παρέμβαση του η δήλωση της πολιτικής, όπως σας είπα, υιοθετείται περίπου στα μέσα της χρονιάς και σε ό,τι αφορά τις αλληλευτικές δυνατότητες εκκινούν από εκεί. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας αυτής όμως είναι μια δημόσια διαβούλευση που γίνεται το καλοκαίρι, η οποία ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε 128 συμβολές από διάφορα εμπλεκόμενα μέλη, από την βιομηχανία, με κυβερνητικούς οργανισμούς, με μονομένους πολίτες και όλες αυτές οι συμβουλές βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας και παρακολουθούνται, εξετάζονται από κοντά από τους συναδέλφους μας και από διάφορα μέλη της ε, διεύθυνσής μας, ούτω ώστε να ετοιμάσουν τις προτάσεις ε, αλληλευτικών δυνατοτήτων. Έχουμε επίσης και κάποιες συστάσεις και συμβουλές από τα διαφορετικά συμβουλευτικά όργανα που συνεργάζονται μαζί μας. Έχουμε λάβει υπόψη μας και όλα αυτά οι συνάδελφοι όταν προετοιμάζουν την πρόταση αλληλευτικών δυνατοτήτων. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ερώτημα και τα σχόλια τη κυρία Μέμορη. σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που θίξατε τα ζητήματα αυτά. Τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Το συγκεκριμένο ερώτημά σα πραγματικά δεν έχω ιδέα τι να σας πω. Και με αυτό λοιπόν ολοκληρώνω. Σε ό,τι αφορά το Brexit, λέει ο πρόεδρο. η... το Ενωμένο Βασίλειο δεν έχει επικυρώσει ακόμη την απόφαση εξόδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η συζήτηση των βιώσιμων ζητημάτων και το, το θέμα της αλίας, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό πιο συγκεκριμένα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά το άρθρο 50 και πίστευω ότι αυτοί είναι αρμόδιοι να απαντήσουν στο ερώτημά σας. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως εγώ, υπάρχει ένα νομοσχέδιο για, τις αλίας, για την αλία αλλά όταν μιλάμε για μέγιστη βιώσιμη απόδοση υπάρχουν και οι δικοί μας στόχοι. Επόμενος γύρος ερωτήσεων. Απλά επιτρέψτε μου να, να σας ρωτήσω ότι πέρα από όλα αυτά τα όμορφα νούμερα που μας παρουσιάσατε, εξαιρετικά νούμερα όπως είπε και ο κύριος Μιγιάν μου, πολύ ενθαρρυντικά. Οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί θα, θα έλεγαν ότι είστε περαισιόδοξοι εσείς στην Επιτροπή και δεν καταφέρνει να λάβει υπόψη όλα τα μη εμπορικά είδη ψαριών. Επομένως, τα 81 τα 81 συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα που παρουσιάζετε δεν είναι και πολύ ενδεικτικά. Άρα, τα νούμερά σας είναι κάπως προσαρμοσμένα στην αισιόδοξη εικόνα που θέλετε να μας παρουσιάσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ καταλαβαίνω και υπό το φως ε, της ε, ανάλυσης που μόλις ακούσαμε, ότι συμφωνούμε πως οι Ευρωπαίοι αλληλείς έχουν ανάγκη από ξεκάθαρους κανόνες και αποτελεσματικούς κανόνες από πλευρά ε, του Ευρωκοινοβουλίου και ολόκληρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μια προσέγγιση αυστηρή, ίση για όλους. Το δεν λειτουργεί και δεν λειτουργεί κυρίως στο τομέα της αλληλείας, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι αγνοούμε την βιοπικιλότητα των θαλασσών μας και τις ιδιαιτερότητες των στόλων μας. Έχω ιδιαίτερα προσφυλές στο θέμα των μικρών αλλιών ε, αυτών της Μεσογείου. Από ό,τι κατάλαβα και η Κομισιόν συμφωνεί στο ότι είναι οι πραγματική ε, φύλακες της θάλασσας. Είναι δηλαδή ένα, ε, ένα οχυρό, ένα φρούριο που προστατεύει τη θάλασσα. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας και όλα αυτά που θα συζητήσουμε σε λίγο στον τριμερή διάλογο για να ενισχύσουμε αυτό του είδους στην μικρή αλία. Εγώ βλέπω από την ανάλυση πως δεν χρησιμοποιείται αρκετά, χρησιμοποιείται λάθος ε, και ε, θα, κάνω ένα παράδειγμα, θα δώσω ένα παράδειγμα. Έχω τα νέα ότι σε μια περιοχή της Νότιας Ιταλίας η περιφέρεια χρησιμοποιεί λάθος 400.000 ε, ευρώ από τα χρήματα των φορολογόμενων για να αναζωογονήσει μια αστική περιοχή ε, ε, ενώ για τους αλληλείς αντίθετα χρειάζεται πάντοτε συγχρηματοδότηση και σε πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά τα 400.000 ενώ ε, για την αστική περιοχή δίνονται τα χρήματα εξ ολοκλήρου. Έπειτα διάβασα ότι 18 από τα 28 κράτη έστειλαν ε, εκθέσεις για τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης. Ποια είναι τα 10 κράτη λοιπόν που δεν έδωσαν ε, τις σχετικές εκθέσεις και με ποιο αιτιολογικό. Έπειτα, εν γέννη βλέπω να δίνεται μεγάλη προσοχή, πολλά γραφήματα ε, για όλες τις θάλασσες, ε, εκτός από την Μεσόγειο. Και αυτό είναι μια περίπτωση που δεν ξέρω, ίσως αργότερα να μας δώσει κάποια συγκεκριμένη έκθεση για την Μεσόγειο θάλασσα. Τέλος, για την απασχόληση. Και εδώ διαβάζω ε, από την Κομισιόν ότι αυξάνεται η απασχόληση. Εγώ δεν έχω δει να γίνεται κάτι τέτοιο και σίγουρα όχι για την αλία μικρή κλίμακα στη Μεσογεία, στη, της Μεσογείου. Ε, γίνεται λόγος και για τη μείωση των τιμών των καυσίμων και αυτό είναι ψευδής ε, είδηση. Τώρα αν μιλήσουμε για την Ιταλία, οι τιμές αυξάνονται. Στην Ιταλία είναι η πιο, έχουμε την πιο ψηλό κόστος για τα καύσιμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και γι' αυτό θα ήθελα εδώ να εμβαθύνουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Απλώς να πούμε ότι στην επόμενη συνεδρίασή μας θα ασχοληθούμε με τη Βόρεια Θάλασσα και με τη Μεσόγειο για να απαντήσουμε σε αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα, αλλά θα δούμε τι έχει να πει η Κομισιόν για το ζήτημα της υποχρέωση εκφόρτωσης. Ευχαριστώ ήδη πολύ προλαλήσαντες. Είπαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εργαστούν με αυτές τις ε, ε, ποστός. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα στην ε, Ανατολική Βαλτική για τον Γάδο είχαμε αύξηση 70% μετά είχαμε 86% μείωση το επόμενο έτος. Μα τι προγραμματισμό να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο και για την Ανατολική Βαλτική. Τώρα έρχεται σύμφωνα με την Κομισιόν μια μείωση κατά 71%. Αυτά προφανώς δεν έχουν σχέση με την αλληλεία, αλλά με άλλους εξωτερικούς ε, παράγοντες. Και εγώ απογοητεύτηκα για το ότι η Κομισιόν χρησιμοποιεί αποκλειστικά αλληλευτικά μέσα. Μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα με τις ποσοστώσεις, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τι γίνεται με τους άλλους παράγοντες, τον ευτροφισμό μέχρι όλα τα άλλα πράγματα που παίζουν τουλάχιστον στη Βαλτική μεγάλο ρόλο παίζει και η κλιματική αλλαγή. Και είναι πολύ βραχυπρόθεσμο να μιλάμε μόνο για αποστώσεις. Ε, αν χρησιμοποιούμε μόνο αυτό το μέσο, ε, τότε τουλάχιστον ε, στη Βαλτική, στη Γερμανία ή μικροί αλείς δεν θα μπορέσουν πλέον να τα ανταποκριθούν. Αναμένω λοιπόν να μας πει η Κομισιόν τι σημαίνει αυτά για το οικοσύστημα και εάν έχουμε πραγματικά τόσο ριζικά μέτρα τα οποία προτείνει, πώς μπορούμε, ε, δηλαδή τι θα κάνουμε, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βοηθούν, δεν μπορούμε να τους ε, το απαγορεύσουμε και να τους αφήσουμε στη μοίρα τους. Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. να έχετε τον λόγο. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την παρουσίαση. Στην Βαλτική Πιστεύω ότι το πολιετές πλάνο ήταν η πρώτη εξέλιξη που έχουμε. Τρία χρόνια μετά έχουμε ε, προβλήματα με τη βιώσιμη αλία. Βλέπουμε ότι τα αποθέματα δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Βλέπουμε ότι γίνεται υπεραλία σε επίπεδα που δεν προτείνονται. Βεβαίως υπάρχουν και άλλοι α, παράγοντες, όπως έλεγε και ο κύριος Μίλαν έχει να κάνει με την, α, με την μόλυνση, η οποία δεν είναι όμως ίδιον της ε, Μεσογείου. Έχει, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και στην Γεωργία, που επηρεάζουν και την ποιότητα του οξυγόνου στην θάλασσα. Μήπως έχετε εξετάσει από κοινού όλες αυτές τις επιπτώσεις μαζί με άλλες γενικές διευθύνσεις με έναν ρεαλιστικό τρόπο. Πιστεύω βεβαίως ότι θα πρέπει να φτάσουμε του, τους στόχους της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. 50, 50 από 59 ήδη αλλιεύονται με βιώσιμο τρόπο. Τι έχουμε να πούμε όμως για τα 59 από τα 200 ήδη. Αν εξετάζουμε α, τα, τα ίδια για το 13. Αυτό που θα ήθελα εγώ να μάθω ήταν πώς, ε, πώς ακριβώς έχουμε προοδεύσει σε ό,τι αφορά μια γενικότερη προσέγγιση. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου λίγο να επιστρέψω σε αυτό το ακαθόδε ζήτημα του, του Brexit. Η συνάδελφος είπε ότι όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, στις 31 Οκτωβρίου όπως μας είπε, πιθανότατα, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάρει πίσω τα ψάρια του. Να ζητήσω εγώ από τη Κομισιόν κατά πόσο υπάρχει ένα συγκεκριμένος μηχανισμός για να μπορούμε να δούμε ποια είναι η εθνικότητα των ψαριών. Μπορεί να μας πει κατά πόσο τα ψάρια έχουν αυτή την ατυχή συνήθεια να πηγαίνουν από το ένα κράτος στο άλλο καμιά φορά να γυρνάνε και πίσω κιόλα. Μπορεί ίσως να μας εγγυηθεί αν το Ηνωμένο Βασίλειο φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται, θα είναι δεσμευμένο από την Σύμβαση των Χωρικών Ιδάτων των Ηνωμένων Εθνών να σεβαστεί και να, να κάνει διαπραγματεύσεις με τις γείτονες χώρες της, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, πάνω σε αυτό που είπε ο πρόεδρος μας τώρα, ο Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι ακόμα θέλει μια συμφωνία και ακόμη διαπραγματεύεται το προσχέδιο αυτής της ε, συμφωνίας που ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. Σε αυτή την περίπτωση ξέρω ότι σε άλλους τομείς που συζητήσαμε και χθε στην ε, Συνταγματική Επιτροπή, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει αναλάβει δράση για να αλλάξει τίποτα. Να υποθέσω ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση και στον τομέα της αλίας. Κάτι θα ξέραμε αν είχαμε αναλάβει δράση. Και επομένως η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι σκοπό να αλλάξει κάτι στο συγκεκριμένο τομέα αν τελικά προχωρήσουμε με τον Brexit. Χαίρομαι που μας διασκεδάζει το Ηνωμένο Βασίλειο γενικά. Ο κύριος Κόρμπετ έκανε κάποια σχόλια. Να επενθυμίσω εγώ ότι δεν υπάρχει κάτι στην ε, ε, συνθήκη που να λέει ότι θα πρέπει να προσδιορίζουμε τι εθνικότητα είναι τα ψάρια. Έχω το κείμενο και ξέρω ότι δεν αναφέρθηκε στα ψάρια. Είμαι σίγουρη που οι ψαράδες, είμαι σίγουρη ότι οι ψαράδες στο Ηνωμένο Βασίλειο θα εκτιμήσουν το χιούμορ του κυρίου Κόρμπετ. Εδώ μιλούσαμε για απόθεμα όμως, δεν μιλούσαμε για κίνηση μεταξύ των χωρικών υδάτων, ελεύθερη κίνηση των ψαριών. Αν δεν έχουμε μια σοβαρή συζήτηση, τότε δεν έχουμε και την ικανότητα να δούμε τις συζητήσεις γίνομαι, γίνονται. Οι ψαράδες, σας το λέω όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε όλη την Ευρώπη θα μας δείχνουν με το δάχτυλο γιατί θα μας κατηγορούν ότι δεν κάναμε την ε, σκληρή δουλειά που να τους επιτρέπει, να τους εξασφαλίζει ότι θα μπορούν να ψαρεύουν στα βρετανικά χωρικά ύδατα. Να ζητήσουμε από την Κομισιόν να απαντήσει, λίγο να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο κύριος Ντεμάτο για τον αριθμό των κρατών μελών που έχουν απαντήσει και δεν έχουν απαντήσει. Ήδη είπαμε ότι το επίπεδο συμμόρφωσης, για να το θέσω ήπια, δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι. Ε, και σε ό,τι αφορά τώρα τα συνολικά επιτρεπόμενα όρια που έχουμε θέσει στην κοινή αλληλευτική πολιτική και την ε, υποχρέωση εκφόρτωσης σε, σε, τι επίπεδο βρισκόμαστε εκεί, σε ό,τι αφορά τι αρχέ βιωσιμότητα κιόλα. Αυτά. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση και την ερώτηση της κυρίας Νταμάτο για την υποχρέωση εκφόρτωσης ε, την στιγμή της ε, δημοσίευσης δεν είχαμε λάβει όλες τις εκθέσεις αλλά τώρα έχουμε λάβει τις ε, περισσότερες βεβαίως οι περίκλειστες χώρες Λουξεμβούργο, Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία δεν χρειάζεται να στείλουμε εκθέσεις Επίσης για την τελευταία ερώτησή σας να επιβεβαιώσω ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν στείλει σχετικές εκθέσεις τους. Για να αναφερθώ σε κάποιες άλλες ερωτήσεις της κυρίας Νταμάτο για το θέμα της απασχόλησης και των μισθών. Έχετε απόλυτο δίκιο για το θέμα της απασχόλησης. Ε, μάλιστα αυτό το οποίο βλέπουμε την τελευταία δεκαετία είναι μείωση της απασχόλησης ε, μεταξύ 2 και 3% το έτος ε, για φυσικούς λόγους, συνταξιοδότηση, γύρανση αλλά και γενικότερη μείωση της χωρητικότητας ε, του στόλου. Βλέπουμε όμως αύξηση των μισθών. Οπότε μειώνεται ε, ο ρυθμός των απασχολούμενων, αλλά αυξάνεται η ποσότητα της απασχόλησης, η ποιότητα, με Οπότε τώρα για τα καύσιμα οι τιμέ ήταν στην κορυφή της ε, κρίσης. Έχουμε εντωμεταξύ μια μείωση των τιμών. Πράγματι η κυρία Νταμάτο έχει δίκιο. Ε, έχει αυξηθεί έτσι η κερδοφορία του όλου, αλλά ξέρουμε ότι γίνονται και δομικές προσαρμογές για να απορροφηθούν οποιασδήποτε άλλαγες ε, στην τιμή ε, της ενέργειας. Ε, τώρα, για τα μη αλληλευτικά μέτρα στη Βαλτική θα τα αναφέρει στην άλλη κυρία Μάγια, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφέρω ε, κάτι το οποίο αναφέρεται σε κάποιες παρεμβάσεις σας. Εμείς είμαστε η Γενική Διεύθυνση Αλίας. Ενώ λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι για το να εξετάζουμε την αλληλεία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό του θαλασσίου περιβάλλοντος είτε μιλάμε για την ποιότητα του νερού, την ποιότητα του πυθμένα, είτε για την κλιματική αλλαγή. Αυτό για το οποίο είμαστε εμείς υπεύθυνοι ως διαχειριστές της αλληλείας είναι οι αλληλευτικές δραστηριότητες. Οπότε, ε, όταν συζητάμε την επιστημονική κοινότητα, στα μοντέλα τους ε, ζητάμε να λαμβάνουν υπόψη και τους μη αλλιευτικούς παράγοντες, κάτι το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι του επιστημονικού τους έργου και όπως εξήγησε ο πρόεδρος όταν η ISS έρχεται εδώ πέρα για να μιλήσει θα σας πει και πόσο δύσκολο είναι να αναπτύξουν συστάσεις για την αλληλεία λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο το οικοσύστημα και τα αλλιευτικά μέτρα. Τέλος. Για το ερώτημα των κυρίων Κόρμπετ και Μοντίθ σας παραπέμπω και πάλι στην Task Force και όχι εξ όσων γνωρίζω στην Κομισιόν δεν ε, εξετάζουμε την εθνικότητα των ψαριών, δεν το παρακολουθεί αυτό κάποιο μοντέλο, αλλά ναι, το Ηνωμένο ε, Βασίλειο έχει κάποιες διεθνείς δεσμεύσεις, όπως ανέφερε ο κύριος Κόρμπετ. Και ε, μετά από αυτά θα δώσω τον λόγο στην Μάγια για να συμπληρώσει τα όσα είπα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα του κυρίου Χέρπστ για την Βαλτική και την δραστική μείωση των ποσοστώσεων. Και μας λέτε πώς θα επιζήσουν. Πράγματι ε, αυτές είναι οι προτάσεις για μείωση 71 και 86% σε Ανατολική και Δυτική Βαλτική. Λοιπόν, ε, θα, το χειρότερο όμως θα είναι εάν καταρρέψουν τα αποθέματα, το οποίο θα συμβεί εάν δεν γίνουν αυτές οι προτάσεις. Και εδώ επανερχόμαστε ακριβώς στα σχέδια τα οποία έχετε αποφασίσει εσείς από κοινού με το Συμβουλίο Υπουργών. Πρέπει να τηρήσουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο είναι μόλις ε, τριών ετών. Οι προτάσεις οποίες ε, κάναμε είναι όλες στο πλαίσιο του σχεδίου. Γιατί προτείνουμε τόσο δραστικές περικοπές. Η ΆΙΣΕΣ είπε καθόλου πλέον αλληλεία στην ε, ρέγγα της ε, Δυτικής Βαλτικής. Αυτή ήταν η επιστημονική συμβουλή μας. χρησιμοποίησαμε το σχέδιο και είδαμε ότι μας δίνει κάποιο περιθώριο και ορίσαμε μια τιμή η οποία είναι στο κάτω όριο της μεγιστής βιώσιμης ε, απόδοσης. Μας δίνεται έτσι η δυνατότητα να λάβουμε ένα επιπλέον μέτρο έτσι ώστε να μπορέσει να ανακάμψει αυτό το είδος. Το ίδιο επίσης ε, και για τον βακαλάο της Δυτικής Βαλτικής. Εάν δεν δράσουμε τώρα θα καταρρεύσει το απόθεμα. Είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε εντελώ και είναι και προ το συμφέρον ακριβώ των μικρών ψαράδων. Βεβαίω είναι σκληρό, βεβαίω είναι δύσκολο, ε, αλλά στον Ατλαντικό παραδείγματο χάρη ε, έχουμε δει καταστάσει όπου ε, καταφέραμε να γυρίσουμε μια δύσκολη κατάσταση κατά 180 μοίρες. Πριν από 10-12 χρόνια είχαμε ένα σχέδιο ανάκαμψης για την ε, χωματίδα αυτή η οποία σήμερα πραγματικά ανθεί. 100.000 ε, τόνους ε, είναι η ετήσια ποσόστοση. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα έχουμε αυτή την ανάκαμψη και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και στη Βαλτική. Και έρχομαι έτσι στο ερώτημα του βουλευτή Ρος και... συγγνώμη. Στο ερώτημά σας και στο ερώτημα του Προέδρου που πάνε λίγο πολύ στην ίδια κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε πως η Κομισιόν έχει κάπως ε, ρόδινα νούμερα και μας είπατε ότι δεν είναι αληθινά. Μιλήσατε, εμείς μιλήσαμε για 59 από 81 και εσείς είπατε για 59 από τα 200. Ε, διαφωνώ. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε την μέγιστη βιώσιμη απόδοση χωρίς τις σχετικές επιστημονικές ε, συμβουλές. Θέλουμε πάρα πολύ να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση σε όλα τα ίδια αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε συμβουλές και για τα 200 είδη. Ε, δεν το έχουμε. Έχουμε μόνο για τα 81. Οπότε ο αριθμός είναι 59 από τα 81 και όπως είπε η συνάδελφος, ε, η οποία είναι η επικεφαλής ε, διαπραγματευτής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αρνητικό ισοζύγιο το οποίο βλέπετε στις διαφανείς είναι κυρίως από τις τρεις χώρες. Εκεί πέρα λοιπόν έχουμε μια, αν μιλήσουμε μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα, 50 από τα 57 ήδη. Κύριε Ρόζα, ανέφερε επίση το σχέδιο τη Βαλτική που είναι μόλι τριών ετών και πράγματι μετά από τρία χρόνια έχουμε μια πολύ διαφορετική κατάσταση στη Βαλτική. Μάλιστα, είχαμε και στο παρελθόν ανάλογε κακέ καταστάσει. Το σχέδιο είναι ένα μέσο για να αλλάξει η κατάσταση, δεν είναι πανάκια. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να λαμβάνονται οι αποφάσεις και αυτό σημαίνει θα πρέπει να γίνονται και οι σωστέ προτάσεις. Ναι, πράγματι τώρα υπάρχει μια αρνητική περιβαλλοντική κατάσταση στην Βαλτική, αλλά δεν χρειάζεται να μειωθούν όλα τα υποθέματα λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων. Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό για το Ανατολικό Πακαλιάρο. Τα υπόλοιπα υποφέρουν από υπεραλίευση. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να μειώσουμε τις ποσοστώσεις. Για ένα χρόνο, για δύο, για περισσότερα, μέχρι η ISIS να μας πει ε, για να ανακάμψουν τα αλλιεύματα, για να αυξήσουμε ξανά στο μέλλον τις ποσοστώσεις. Τώρα πώς θα δούμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει προφανώς να δούμε το θέμα της ε, υπερθέμας του πλανήτη, σαφώς πιο βιώσιμη γεωργία Αλλά εντάξει, δεν έχει νόημα να λέμε ότι το ψάρι αυτό δεν πεθαίνει λόγω αλληλεία, πεθαίνει για άλλου λόγου. Άρα δεν θα λάβω αλληλευτικά μέτρα. Πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση. Ελπίζω να απάντησα σε όλε τις ερωτήσει. Εάν όχι, ε, παρακαλώ να μου το επιθυμήσετε. Λαμβάνεται υπόψη ε, επίσης ε, την υπόθεση ότι θα συνεχίσει να υπάρχει απαγόρευση απόρριψης, ότι υπάρχει υποχρέωση εκφόρτωσης και υπάρχει και το ερώτημα της κυρίας Ρους ότι εντάξει 81 ήδη έχουν αξιολογηθεί επιστημονικά, πότε θα αξιολογηθούν και άλλα. Um, yes, thank Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με τις ε, ποσοστώσεις και τις επιπλέον ποσοστώσεις ε, που έχουν τα κράτη-μέλη μέσω της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Εμείς είπαμε ότι όταν αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η υποχρέωση και θα υποχρεώνονται να φέρουν όλα τα αλλιεύματα στην νυχτιόσκαλα οι ψαράδες ε, θα ξεκινήσουμε με το να τους δίνουμε τις προστώσεις για τα αποθέματα τα οποία πετούσαν ε, στο παρελθόν στη θάλασσα. Τώρα, δικαίως ε, λέτε και το επεσήμανε και η ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν γίνεται σεβαστή αυτή η υποχρέωση παντού. Επ' αυτού το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη θα βελτιώσουν τους ελέγχους ε, στα σκάφη γιατί μόνο έτσι θα γίνει. Και ακριβώς ε, έλαβαν τις ε, ποστώσεις για να φέρουν τα ψάρια όλα πίσω στην εκτός και αυτό αναμένουμε να γίνει. Επίσης νομίζω ότι είπατε κάτι πολύ σημαντικό όταν είπατε πότε θα έχουμε ε, επιστημονικές συμβουλές για περισσότερα Εμεί Εμείς ε, το θέλουμε για όλα. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα ερευνητικά Ινστιτούτα των Καρτών Μελών και το ΆΕΣΙΣ να αφορούν όλα τα αποθέματα που είναι στα σχέδια και έχουμε πάει πλέον σε κάποιες προληπτικές ε, συμβουλές. Σε κάποια άλλα έχουμε συμβουλές για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζονται ερευνητέ στα εθνικά ερευνητικά Ινστιτούτο για να αναπτύξουν τα μοντέλα. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα αποθέματα ε, στον Ατλαντικό. Ε, στον Ατλαντικό και στην, ε, στον Βυσκαϊκό κόλπο. Το θέμα μας λοιπόν είναι με τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν έχουν αρκετού ερευνητέ και αρκετού πόρου γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία για να καταρτήσουμε ένα μοντέλο για την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ελπίζουμε λοιπόν να αυξηθούν τα στοιχεία αυτά που λαμβάνουμε από τον ΆΙΣΕΣ Έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. αλλά απέχουμε ακόμα πολύ από τα 200 είδη που σωστά αναφέρθηκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ, ναι, συγγνώμη, κύριε Μοντίθ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την υπομονή σας. Στο πνεύμα αυτό της ε, συναδελφικότητας ε, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση και πρόταση. Είχα θέσει το θέμα της αποζημίωσης για τους ψαράδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit και στην συνάδελφους εδώ έκανε κάποιες ερωτήσεις για τα αλλιεύματα. Ε, λαμβάνουμε αποφάσεις ε, μονοσύλλαβες θα έλεγα, χωρίς λεπτομέρειες, έτσι αναγκαζόμαστε να κάνουμε γραπτές ερωτήσεις, μας παραπέμπουν στην Task Force. Θα ήθελα να προτείνω σε μία από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας ε, πριν το Brexit που ίσως γίνει στις 31 να καλέσουμε την Task Force εδώ πέρα έτσι ώστε όλοι μας να κάνουμε ερωτήσεις. Τι γίνεται για να βοηθήσουμε τους ψαράδες ε, μετά το Brexit. Είτε υπάρχει συμφωνία είτε όχι. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό για όλους μας ε, και νομίζω ε, θα μας βοηθήσει και για να υπάρχει διαφάνεια αντί να μας λένε δεν είναι δικιά μου ευθύνη και δεν ξέρω τι να πω. Σας ευχαριστώ κύριε Μοντίθ. Ε, συμφωνούμε και εγώ θα ήθελα να βάλω κάτι στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Οπότε θα έχω και εγώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση για την υπεραλίευση. Κύριε Κέσνερ. Και οι δυο σας έχετε πει ότι δεν πρέπει να υπεραλείβουμε, αλλά δεν έχει νόημα να είμαστε ευγενικοί βραχυπρόθεσμα, γιατί ε, έτσι μακροπρόθεσμα θα εξαφανιστεί ο κλάδος. Ή όχι και τόσο μακροπρόθεσμα. Ε, και όμως υπάρχουν κάποιες στιγμές ε, που γίνονται οι συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου και η Κομισιόν κάνει κάποιες συστάσεις για ποσοστώσεις πάνω από την Επιστημονική Συμβουλή. Γιατί το κάνετε αυτό. γιατί δεν ακολουθείτε πάντα τις επιστημονικές συμβουλές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα την αίσθηση ότι θα γινόταν αυτή η ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που γίνεται συχνά. Πάντα ε, λαμβάνουμε επιστημονικές α, ε, συμβουλές προκατακτικές για τα είδη πλην των 81 ειδών. Θα ήθελα να αναφερθώ στον επιστήμονα της ISIS, ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκεκριμένα, όταν ε, δέχτηκε ακριβώς την ίδια ερώτηση σε ένα συνέδριο και εκεί ένας ομιλητής είπε ότι στο 44% των περιπτώσεων τα συνολικά επιτρεπτά λιεύματα είναι πάνω από την Επιστημονική Συμβουλή. Και η απάντησή του ήταν ότι η αριθμοί αυτή είναι λάθος γιατί ε, περιλαμβάνουν ε, δεδομένα από όλα τα αποθέματα. Αυτό, αυτή τη φράση είπε. Δηλαδή ε, ισχύει αυτό το οποίο είπατε, ναι, η Κομισιόν θα μπορούσε να λάβει αυτήν την συμβουλή που είναι φτωχή σε δεδομένα. Ο για τα δύο είδη που ανέφερα πριν, αν ε, κάποιος ενδιαφέρεται για τον ε, μπακαλιάρο αυτόν. Εδώ πέρα μιλάμε για μια επιστημονική συμβουλή η οποία δεν έχει επαρκή δεδομένα. Ε, και έχουμε ένα είδος το οποίο είναι στόχευμένο σύμφωνα με το σχέδιο. Τι λέει η συμβουλή, απλοποιώ τώρα εδώ πέρα, λέει ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ξέρουμε ότι είναι πολύ υψηλό το συνολικό επιτρεπτό αλίευμα γιατί βλέπουμε ότι οι ψαράδες ε, ξεφορτώνουν μόνο 40% του συνολικού αλίευματος. Επίσης λέει η Συμβουλή ότι δεν μπορούμε να δώσουμε προφορίες εάν είναι πολύ υψηλή η αλευτική πίεση για το αν εντάξει η βιομάζα. Δεν μπορούμε, να πούμε, πώς η βιομάζα υπάρχει στη θάλασσα. Σας λέω αυτές τις πληροφορίες για να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν ε, διάφορα είδη ποιότητα επιστημονική συμβουλή. Εντάξει, κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά αυτό εξαρτάται από τα στοιχεία που δίνουν τα κράτη-μέλη και τα εθνικά ερευνητικά κέντρα. Εάν δεν γίνει η δουλειά στην Ιρλανδία και στη Γαλλία, δεν μπορούν να κάνουν περισσότερα και στο ISIS. Οπότε για να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο που κάθε χρόνο μας λένε ναι, τι γίνεται με όλα τα υπόλοιπα, δεν ακολουθείτε τις επιστημονικές συμβουλές. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα όλα τα είδη στόχο και να έχουμε επιστημονικές ε, συμβουλές. Και σας πόσχομαι ότι τη στιγμή που θα έχουμε επιστημονική συμβουλή και για το συγκεκριμένο ε, είδος θα προτείνουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό και ούτε ένα τόνο παραπάνω. Αυτό έχουμε κάνει σε όλα τα είδη για τα οποία έχουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ελπίζω να απάντησα. Ευχαριστώ, δεν βλέπω κάποιον άλλο να θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και τις δυο σας. Βέβαια, εντάξει, μπορεί η Επιτροπή να ε, ασκήσει κάποιες ε, κριτικές και μπορεί να πούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες θάλασσες και αλλιεύματα που δεν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά Όσοι μιλάμε με ψαράδες μας λένε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι 15-20 χρόνια στις περισσότερες θάλασσες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπάθειές σα. Thank you very much. So, item 9. Study on engine. Μελέτη για την υποδύναμη των ε, κινητήρων. Μη φεύγετε κύριε Άλλαρντ. Ακούγεται βαρετό αλλά δεν είναι. Ζήτησα από την Επιτροπή να μας υποβάλει την πρόσφατη μελέτη για την υποδύναμη των ε, κινητήρων όπως ξέρετε, η υποδύναμη των κινητήρων των αλληλευτικών σκαφών είναι ένα από τα μέσα ελέγχου της αλληλευτικής προσπάθειας και στη Μεσόγειο για να καθοριστεί ο, επίσης ο, το μέγεθος του Ευρωπαϊκού Αλληλευτικού στόλου και έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αλλιεύουμε βιώσιμα. Και η επαλήθευση αυτή είναι σημαντικό κομμάτι της συζήτησης στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον κανονισμό περί ελέγχου και τις σχετικές εφαρμοστικές διατάξεις. Όπως γνωρίζουμε θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του κανονισμού περιελέγχου και θα μεριμνήσουμε με τις τροπολογίες μας να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ακρίβεια της πιστοποιημένης ε, υποδύναμης. Το θέμα είναι η ισχύουσα κατάσταση είναι ικανοποιητική ή συζητείται πάντοτε κατά πόσο είναι ακριβής η ε, δυνατότητα των καταμετρημένη δυνατότητα του λευτικού στόλου. Δώσω το λόγο λοιπόν στον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν για να μας, ε, στην εκπρόσωπο της Κομισιόν για να μας καθοδηγήσει και να μας εξηγήσει αυτή τη μελέτη. Ε, κυρία Αρένα, καλησπέρα σας. Ε, πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα πορίσματα αυτής της μελέτης, η οποία πρόσφατα ολοκληρώθηκε, δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, οπότε είναι φρέσκια, τα αποτελέσματα είναι ακόμα πολύ πρόσφατα και η συνέχεια αυτής της μελέτης από πλευράς της Κομισιόν ε, δίνεται ήδη. Πριν να προχωρήσουμε στις λεπτομέρειες της μελέτης, θα ήθελα να σας δώσω το πλαίσιο για αυτήν. για την υποδύναμη των ε, μηχανών. Σωστά στην εισηγωγή σας μιλήσατε για αλληλευτικές δυνατότητες και η δυνατότητα και τα όρια της ορίζονται από την κοινή αλληλευτική πολιτική Επίσης ορίζονται απαιτήσεις για τα σχέδια εισόδου-εξόδου, δηλαδή πώς η αλευτική δυνατότητα μπορεί να μπει στον αλευτικό στόλο ενός κράτους μέλους και πώς η αλευτική δυνατότητα πρέπει να ε, καταστραφεί. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο, σε περίπτωση που γίνεται χρήση ενωτικών χρημάτων, δε, τότε η αλευτική δυνατότητα που καταστρέφεται δεν θα πρέπει να τα καταστρέφεται από νέα ε, δυνατότητα. Έπειτα υπάρχουν διάφορα προγράμματα που λειτουργούν στην Ένωση υπάρχουν τα καθεστώτα αλληλευτικής προσπάθειας τα οποία ορίζονται σε διάφορα πολιετή σχέδια. Εδώ αναφέρω το πολιετές πρόγραμμα για τη Βόρεια Θάλασσα αλλά και τα πολιετή προγράμματα για τη Δυτική ε, Μεσόγειο. Και τέλος, στο τεχνικά μέτρα, ε, ε, το νέο, ο νέος κανονισμός ε, περί τεχνικών μέτρων υιοθετήθηκε επίση πρόσφατα, περιλαμβάνονται διάφοροι περιορισμοί όσον αφορά τα σκάφη πέρα από τα 221 κιλοβάτ για διάφορες περιοχές, βόρεια θάλασσα, βόρειο-δυτικά ύδατα και βαλτική θάλασσα. Στις ε, διατάξεις περιαλίες περιλαμβάνονται και διάφορες διατάξεις όσον αφορά την αλευτική δυνατότητα και πιο συγκεκριμένα για την υποδύναμη των ε, μηχανών. Πράγμα που μας φέρνει στο επόμενο σημείο, δηλαδή στο γεγονός ότι αυτοί οι διατάξεις και εφαρμογή τους θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγχονται και γι' αυτό το λόγο το 2009 τροποποιήθηκε ο κανονισμός περί ελέγχων και εισήχθησαν διάφορα άρθρα για τον έλεγχο των αλληλευτικών δυνατοτήτων και την υποδύναμη των μηχανών που συμπληρώθηκαν από εφαρμοστικούς κανόνες που υιοθετήθηκαν από την Κομισιόν το 2011. Συνοπτικά λοιπόν τι σημαίνει έλεγχος της υποδύναμης σήμερα. Σημαίνει πως τα κράτη-μέλη πρώτον πρέπει να πιστοποιούν την ε, υποδύναμη σε κιλοβάτ και να διευκρινίζουν αυτή την υποδύναμη στην άδεια. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο νεολόγιο του κράτους και στο ενωτικό νεολόγιο. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν υπερβαίνεται αυτό το όριο του στόλου, ε, το πιστοποιημένο ε, και το αδειοδοτημένο. Πώς γίνεται αυτό. Κάνουν, ε, φτιάχνουν ένα σχέδιο δειγματοληψίας για να επαληθεύσουν ε, την υποδύναμη των σκαφών. Εντοπίζουν ας πούμε τα λευτικά σκάφη, για παράδειγμα αυτά που έχουν πολύ μεγάλα τονάζ και μικρή μηχανή, φαίνεται να έχουν μικρή μηχανή, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτά τα σκάφη χρησιμοποιούν όλη τους την υποδύναμη για να κινηθούν και δεν θα είχαν πια άλλη ε, υποδύναμη για να μπορέσουν να αλλιεύσουν, για να λειτουργήσουν τα ε, μηχανήματα. Ε, αυτά τα ίδια λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διεξάγουν πραγματικούς ελέγχους της υποδύναμης επιτόπου και πλέον να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, εφόσον εντοπίσουν σοβαρές παραβάσεις γιατί μία λαθασμένη ψευδής δήλωση ε, σχετικά με την υποδύναμη του κινητήρα θεωρείται σοβαρή παράβαση. Στο παρελθόν η Κομισιόν ε, είχε διαπιστώσει πως δεν ε, γινόταν επαρκής ε, εφαρμογή των δειγματοληπτικών σχεδίων. Υπήρχαν πολλές παραβάσεις και είχαμε λάβει διάφορες καταγγελίες στη διάρκεια των ετών και γι' αυτό αποφασίστηκε η εκπόνηση της μελέτης αυτή στη διάρκεια του 2018 ώστε να ε, επαληθευθεί η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Να δούμε δηλαδή ποια ήταν η πραγματική κατάσταση στα κράτη-μέλη, γιατί είναι σαφές ότι χωρίς αποτελεσματικό έλεγχο υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχουν υπερβάσεις των αλληλευτικών δυνατοτήτων και αυτό θα οδηγούσε σε έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στην ε, αλληλευτική δυνατότητα και την αλληλευτική ε, ευκαιρία ε, και άρα την θέση σε κίνδυνο της ίδιας της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θέλαμε λοιπόν να εντοπίσουμε ποιες ενέργειες είχαν, σε ποιες ενέργειες είχαν προβεί τα κρατημέλη, συγκεκριμένα να δοκιμάσουμε αρκετούς κινητήρες και το κάναμε αυτό σε ένα δείγμα σκαφών, αλλά θέλαμε θέλαμε να δούμε, να εξετάσουμε και το τι ακριβώς γίνεται να εντοπίσουμε τις καλές πρακτικές για τη δειγματοληπτικό έλεγχο των ε, μηχανών, των κινητήρων και ποιες ήταν οι καλύτερες πρακτικές για τον έλεγχο της ε, αληπτικής προσπάθειας ε, του εκάστοτε στόλου. Ε, το εύρος της μελέτης ήταν αρκετά μεγάλο. Ε, φέραμε να καλύψουμε 15 κρατημέλη σε μια περίοδο 1,5 έτους. Ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2018 και ολοκληρώσαμε τον Ιούνιο φέτος. Ε, μελέτη έγινε από δύο ομίλους, δύο εταιριών και δύο υπεργολαβών, των οποίων ηγείται μια Ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται σε δοκιμές κινητήρων. Έγιναν διάφορες ε, συνεδριάσεις που διοργανώθηκαν με τις ε, κρατικές αρχές των ε, κρατών μελών και έγιναν και ευνίδιοι έλεγχοι ε, της ε, υποδύναμης των ε, κινητήρων σε 68 κράτη, σε 14 κράτη-μέλη. Σε ένα μόνο κράτος μέλος δεν κατέστη δυνατόν να κάνουμε τέτοιον ευνίδιο έλεγχο. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η πραγματική αυτή επιτόπιοι έλεγχοι έγιναν ευνίδια. Δηλαδή, οι αρχές γνώριζαν ότι θα γίνουν έλεγχοι, αλλά ο εντοπισμό του σκάφους ε, γινόταν τελευταία στιγμή και το ίδιο το λευτικό σκάφο δεν γνώριζε ότι πρόκειται να υποστεί σε έλεγχο ε, ε, να υποστεί έλεγχο. Έγιναν λοιπόν έλεγχοι σε διάφορα σκάφη. Μπορείτε να δείτε στον κατάλογο τα είδη των σκαφών που ελέγξαμε και ο αριθμός των σκαφών ήταν, που ελέγχθηκαν ήταν αντίστοιχος με το μέγεθος του στόλου του κάθε κράτους μέλους. Τώρα, ποια ήταν τα πορίσματα. Τα πορίσματα διόλου θετικά πρέπει να σας πω. Μάλιστα, πολύ ανησυχητικά είναι, διότι εδώ βλέπετε συνοπτικά το κόκκινο κομμάτι εδώ του σχήματος, το κόκκινο και το πράσινο δείχνουν ότι 51% των σκαφών που ελέγχθηκαν δεν ήταν σύμμορφα προς τους κανόνες. Δηλαδή πάνω από 100% της πιστοποιημένης υποδύναμης είχαν. Αν περιλάβουμε και το υπόλοιπο 60%, 60% ε, το κόκκινο και το πράσινο, βλέπουμε ότι το 67% των σκαφών που ελέγχθηκαν είτε δεν ήταν ε, σύμμορφα, είτε υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Μόνο το 1 τρίτο δηλαδή του δείγματος τελικά ε, ήταν ε, πλήρως σύμμορφο με τους κανονισμούς. Μόνο το 1 τρίτο των σκαφών που ελέγχθηκαν. Αν αυτό το μεταφράσουμε και από την πλευρά των αλλιέων, αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι ανησυχητικά μόνο από την άποψη της κοινή ε, αλληλευτικής πολιτικής, πολιτικής, αλλά και για τους ε, αλληλείς που συμμορφώνονται προς τους κανόνες. Αυτό μας οδηγεί στο επίπεδο συμμόρφωσης. Συνοπτικά, η μη συμμόρφωση ε, διαπιστώθηκε σε 10 από τα 14 κράτη-μέλη και εν γέννη σε κάθε στόλο που ελέγξαμε. Δεν υπήρξε κανένα κομμάτι δηλαδή του ευρωπαϊκού στόλου το οποίο να ήταν απόλυτα πράσινο, απόλυτα σύμμορφο. Και το, το ποσοστό και το μέγεθος της μη συμμόρφωσης είναι πραγματικά ανησυχητικό, άρα λοιπόν πρέπει να, να, να προβούμε σε ενέργειες. Επίση, σημαντικά αποτελέσματα είχαμε για τη διαδικασία πιστοποίηση, που είναι το πρώτο βήμα ε, για τον έλεγχο τη υποδύναμη. Ε, το, το, το πόρισμα ε, τη μελέτη είναι ότι τα ισχύοντα συστήματα πιστοποίηση δεν ανταποκρίνονται στο στόχο γιατί εάν κανείς πιστοποιήσει έναν κινητήρα, έπειτα στη συνέχεια με τον επιτόπο έλεγχο θα ανέμενε κανείς το ίδιο αποτέλεσμα που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, πράγμα που δεν συμβαίνει. Επίσης είδαμε, διαπιστώσαμε ότι τα, ε, το έργο της πιστοποίησης ανατίθεται από τις αρμόδιες αρχές σε κάποια άλλα όργανα και συχνά δεν υπάρχει αναντιστοιχεία. Τα καλά νέα σε κάποια κρατημέλη γίνονται συστηματικοί έλεγχοι όσον αφορά την πιστοποίηση. Τι σημαίνει αυτό, ότι πριν τη χορήγηση ενός πιστοποιητικού κάνουν πραγματικό επιτόπιο έλεγχο. αλλά στα υπόλοιπα κράτη-μέλη η πιστοποίηση δίνεται χωρίς επιτόπιο έλεγχο, μόνο δηλαδή μέσω του ελέγχου γράφων, πράγμα που δεν αρκεί. Το σύστημα πιστοποίησης ε, που εφαρμόζεται από τις αρμόδιες ε, ε, αρχές. Επίσης είναι λοιπές. Κάποιες φορές δεν γίνεται καθόλου συστηματικά. Σε άλλα κράτη-μέλη ε, γίνονται αναλύσεις αποτελεσμάτων μόνο μια φορά στα 10 χρόνια. Ε, μόνο τρία κατημέλη έκαναν επιτόπιους ελέγχους στους κινητήρες. στο ένα υπό το νομικό πλαίσιο του κανονισμού περιλέγχου Τρία κράτη-μέλη από τα 15 ε, ε, αξιολογούν συστηματικά τα πιστοποιητικά. Συμπέρασμα είναι ότι ακόμα και όταν εφαρμόζεται το σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό, γιατί σε κάθε περίπτωση υπήρχε πολύ ψηλό ποσοστό μη συμμόρφωσης των ε, κινητήρων που ελέγχθηκαν μέσω αυτής της μελέτης. Πέρα από αυτά τα αποτελέσματα, λοιπόν, οδηγηθήκαμε, μάλλον με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οδηγηθήκαμε σε συστάσεις και εδώ τι συνοψίζουμε. Η πρώτη αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης που πρέπει σίγουρα να βελτιωθεί, αλλά και να εναρμονιστεί. Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση της νομοθεσίας, για παράδειγμα εγκατάσταση της λιγότερο ισχυρής, του λιγότερου ισχυρού κινητήρα που είναι διαθέσιμος να ορίσουμε την ε, την αποκατηγοριοποίηση ε, την διεύρυνση των απαιτήσεων αλλά και την ένταξη, την εισαγωγή μάλλον νέων και, και, στα, και στάνταρ διαδικασιών για την ε, επαλήθευση και τον έλεγχο. Προτείνουμε διαρκή παρακολούθηση των ε, κινητήρων. Αυτό θεωρήθηκε από τους μελετητές ως πολύ καλό εργαλείο, αλλά όχι για τα μικρά σκάφη βέβαια. Ε, θα ήταν ένα εργαλείο που θα μπορούσε να ε, ελέγξει κατά προτεραιότητα τα σκάφη υψηλού κινδύνου ή τα σκάφη όπου οι κινητήρες δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι. Υπάρχουν και άλλα ε, εργαλεία, αλλά εδώ νομίζω θα μπούμε σε πολύ τεχνικές λεπτομέρειες που δεν θα ήθελα να σας κουράσω με αυτές για την ώρα. Πέρα από αυτές τις βασικές συστάσεις θα είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις λόγω του ανεπαρκούς ελέγχου της υποδύναμης των κινητήρων και οι επιπτώσεις αυτές αφορούν τα σχέδια εισόδου και εξόδου και την στήριξη από το Ταμείο και για αυτά τα θέματα θα ήθελα σύντομα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Ελίζα. Ευχαριστώ, Φρανσέσκα. Δύο πράγματα θέλω να πω για το σύστημα εισόδου-εξόδου και για το ταμείο. Παράλληλα με την έρευνα επαλήθευση ισχύ κινητήρα, κάναμε και μια αξιολόγηση του συστήματο εισοδου εισόδου-εξόδου. Και τα δύο μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Το σύστημα εισόδου-εξόδου λέει ότι αν πάρει κάποιος επιδότηση, δημοσιοεπιδότηση, για να σταματήσει να χρησιμοποιεί ένα σκάφος, αλευτικό σκάφος, θα πρέπει να αφαιρεθεί και η δυνατότητα από τα ανώτατα όρια δυνατότητας που διαθέτει κάθε κράτος μέλος. Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να ελέγχουμε την ε, δυνατότητα να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε σύμφωνα με το στόλο. Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στα κράτη-μέλη, ένα ευέλικτο εργαλείο που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χειρίζονται τους στόλους που έχουν. Το, το, η επαλήθευση της ισχύς του κινητήρα είναι πολύ σημαντικό για το συγκεκριμένο σύστημα, γιατί για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η δυνατότητα του στόλου, πρέπει να μπορούμε να καθορίσουμε και το μέγεθος του σκάφους, είτε μέσω ΆΣ είτε μέσω της ισχύς του κινητήρα. Και αυτό που η έρευνα της αξιολόγησης μας είπε είναι ότι είναι λειτουργικό το μέτρο αυτό, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν το εφαρμόζουν αποτελεσματικά. Επομένως υπάρχει μία συζήτηση σε όσο αφορά τη δυνατότητα και βασικό σημείο της δυνατότητας είναι αυτό το σύστημα εισόδου-εξόδου η μη αποτελεσματικότητα του συστήματος δεν οφείλεται στα ανώτατα όρια ή στον τρόπο που έχει οριστεί, αλλά στην μη σωστή εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη. Και γιατί το λέμε, γιατί συνδέεται με το Ταμείο, με το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Αυτή τη στιγμή στο Ταμείο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πόρους α, για να αυξήσουμε τη δυνατότητα ενός σκάφους μέσω χορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα βάλουμε στην πρόταση της Κομισιόν για μετά το 2020 για το τιμίο. Αλλά αυτή τη στιγμή που λαμβάνει χώρα η διαδικασία συν οι συνομοθέτες έχουν αποφασίσει κατά πώς φαίνεται ότι το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει μία σειρά από επενδύσεις ενδυνάμωσης της δυνατότητας, περιλαμβανομένου και της αντικατάστασης των κινητήρων, χωρίς να γίνεται προηγουμένως επαλήθευση και χωρίς να υπάρξει υποχρεωτική οδηγία μείωσης της ισχύς του κινητήρα. Πιστεύω ότι αυτό που δείχνει η έρευνα επαλήθευσης ισχύς ε, του κινητήρα είναι ότι αν δεν εφαρμόσουμε τους κατάλληλους ελέγχους, η διαχείριση της δυνατότητας, η χρήση του ταμείου δεν γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνονται. Αυτό απλά θέλαμε να προσθέσουμε εμείς εδώ, επιπλέον σε αυτά που είπε η Φρανσέσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. And with this we can move uh, και μπορούμε τώρα να περάσουμε στην τελευταία διαφάνεια που έχει στόχο να σας παρουσιάσει ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε. Όπως είπα στην αρχή της παρουσίασής μου, θα ξεκινήσουμε μια σειρά από δράσεις, ακόλουθες δράσεις για τα 14 κάτι μέλη όπου κάναμε δοκιμές. θα ζητήσουμε επαλήθευση εκεί όπου δεν υπήρχαν, εκεί όπου διαπιστώσαμε ε, μη συμμορφούμενα περιστατικά, να δούμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δράση. Επίσης, θα επαληθεύσουμε ότι τα κράτη-μέλη όπου διαπιστώσαμε ελλείψεις στα πιλωτικά προγράμματα θα βελτιώσουν το σύστημα ελέγχου τους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα αυτά ε, γύρουν ανησυχίες για το γενικό επίπεδο συμμόρφωσης και στα υπόλοιπα που δεν κάλυψε η μελέτη. Ο λόγος ήταν ο περιορισμένος προπολογισμό που είχαμε εκείνη την εποχή, επομένως έπρεπε να επιλέξουμε. Η Επιτροπή τώρα θα ξεκινήσει μια έρευνα για να μπορέσει να έχει ανάλογες πληροφορίες και από τα κράτη-μέλη που δεν εξετάσαμε, τόσο ώστε να έχουμε μια γενικότερη αξιολόγηση. Τέλος, είναι σαφές ότι η έκθεση αυτή θα είναι πολύ χρήσιμη για να ενημερώσει όλες αυτές τις συζητήσεις για τον κανονισμό που σκοπεύουμε να εκδώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Για να δούμε το γενικό πλαίσιο. Αυτό που λέμε είναι κατά πόσο η αλληλευτική προσπάθεια έχει στόχο να διατηρήσει την βιωσιμότητα, κυρίως εκεί που χρησιμοποιούνται ποσοστώσεις ΤΑΚ. Αναφερόμαστε στην Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο. Για, για πόσα ακόμη κράτη-μέλη μιλάμε εδώ. Πώς ακόμη κρατημέλη εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Well, Όπως είπα και στην αρχή της ε, παρουσιασής μου, δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη της Μεσογείου. Υπάρχουν όρια δυνατοτήτων που αφορούν όλα τα κρατη στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Επομένως υπάρχει ένα ανώτατο όριο, το οποίο αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Και όπως σας εξήγησε και η συνάδελφός μου η Ελίζα, υπάρχει το καθεστώς εισόδου-εξόδου και οι διατάξεις του Ταμείου, που είναι πολύ σχετικές με την ισχύ του κινητήρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αλευτικές προσπάθειες, αυτή ήταν η ερώτησή σας. Είναι αλήθεια ότι το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όταν μιλάμε για τάκ και για ποσοστώσεις, δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα αλευτικής προσπάθειας. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν διατάξεις για περιορισμούς αλευτικής προσπάθειας στην ε, Βόρεια Θάλασσα αλλά και στα Δυτικά Ήδατα αλλά και ε, τεχνικά μέτρα και για τη Βαλτική. Επομένως, όλα τα κρατη ε, αφορά όλα τα κρατη που ασκούν αλληλευτική δραστηριότητα σε όλα αυτά τα, σε όλα αυτά τα μέρη που αναφέραμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο θα έχουν την δυνατότητα τα κράτη-μέλη αυτά να, έχουν ε, εκθέσεις. Υπάρχουν ε, πολλά, πολλά στρώματα σε αυτές τις μελέτες. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα άτομα, αυτούς που χειρίζονται τα σκάφη. Η Κομισιόν λέει ότι υπήρχαν ε, δευτερεύοντα στοιχεία όπου οι, οι χρήστες που δεν υπερέβησαν τα όρια κινητήρε του, μπορεί και να, κάπως να, να, πείραξαν τα αποτελέσματα, ούτω ώστε να φανεί ότι οι κινητήρε είχαν χαμηλότερη ισχύ. Και μετά υπάρχει και το δεύτερο ζήτημα, που έχει να κάνει με τους κατασκευαστές, με τους προμηθευτές των κινητήρων και των σκαφών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στα περισσότερα κράτη-μέλη μπορούν ε, οι ψαράδες να εγκαταστήσουν μια μηχανή που έχει μια ισχύ πολύ μεγαλύτερη, αρκεί να υπάρχει μια δήλωση που λέει ότι η ισχύ του κινητήρα είναι όσο αναγράφεται στην άδεια. Και αυτή την ε, πιστοποίηση μπορεί να τη δώσει ο κατασκευαστής. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι παράνομο. Και βεβαίως υπάρχει και το όλο ζήτημα των ίδιων των κρατών μελών που δεν κάνουν τίποτα για να εφαρμόσουν τις διατάξεις της νομοθεσίας που είναι σε ισχύ ελάχιστες επιθεωρήσεις και σε πολλές περιπτώσεις καθόλου επιθεωρήσεις. και με τον ένα τρόπο ή τον άλλο είναι εντελώ ανεπαρκή η έλεγχη εντελω ανεπαρκης η Αυτό που θα έλεγα λοιπόν εγώ τώρα, αυτό που θα πρότεινα, η βάση των αληφτικών μας πολιτικών ε, δεν, δεν είναι ε, ε, πραγματική. Με άλλα λόγια, Πώς μπορούμε να χτίσουμε μια διώσιμη ελευτική πολιτική όταν η βάση μας είναι διεφθαρμένη. Δεν ξέρω αν τα κράτη-μέλη έχουν να πούν κάτι πάνω σε αυτό, αν έχουν κάποια σχόλια. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή που μας έκανε αυτή την ε, ε, παρουσίαση. Είναι ένα θέμα πολύ πολύ τεχνικό και είμαι βέβαιος ότι όπως και οι συνάδελφοι θα σκέφτονται ότι με το που γυρίσαμε από τις διακοπές το να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια έκθεση και να τη διαβάσουμε και να τη μελετήσουμε είναι καταστροφικό. Είναι μια ε, ε, έκθεση πολύ περίπλοκη και τεχνική ακόμα περισσότερο για έναν ναυπηγό παρά για έναν πολιτικό που έρχεται από τον κόσμο του δικαίου. Ε, αυτό που καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα είναι ότι δεν τηρείται η, οδηγία, ο κανονισμός. Αυτό το καταλάβαμε πολύ καλά. Τώρα, πριν από ένα χρόνο επέβαλε την αναθεώρηση του κανονισμού η Κομισιόν και προβλεπόταν για αυτό το είδος ε, παράβαση για όσον αφορά την υποδύναμη του κινητήρα έναν ε, μηχανισμό παρακολούθησης μόνιμο. Βλέπω όμως ότι και με βάση αυτή εδώ τη μελέτη ε, επιμένει σε αυτή την πρόταση. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η θέση της εκπροσώπου της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν, έλεγε, δεν λέει ότι είναι το καλύτερο σύστημα, λέει για δαπάνε αν θυμάμαι καλά, για ένα κόστο ανάμεσα στα 10 και στα 15.000 ευρώ ανά σκάφο το να εγκατασταθεί δηλαδή τέτοιο σύστημα μόνιμης παρακολουθήση. Επίση αυτό το σύστημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα μικρά σκάφη και για ορισμένα σκάφη που είναι ηλεκτρικά, είναι μειχτά, δηλαδή χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό και ντίζελ, δεν μπορεί καν να τοποθετηθεί. Δεν ξέρω ακριβώς δηλαδή αν η Κομισιόν σκοπεύει να κάνει κάνει νέα δήλωση και αν έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες. Εγώ αυτά πάνω κάτω μπόρεσα να καταλάβω. Και θα ήθελα η Κομισιόν να μας πει σε ποιο βαθμό αυτή η μελέτη που μόλις ε, εκδόθηκε μπορεί να αλλάξει την οπτική της για τον ε, κανονισμό ελέγχου. Επίσης θα ήθελα να ξέρω τι είναι, ε, ποια είναι η γνώμη των κρατών μελών, γιατί στην ουσία τον έλεγχο τα κάτι μελη πρέπει να τον ασκήσουν. Επίσης, δεν ξέρω αν ε, το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με αλλαγή των κανόνων, γιατί δεν είναι θέμα κανόνων. Ε, θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν και να μπορούν να ελεγχθούν. Ε, αυτοί οι κινητήρες, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να έχουν μέσα τους μηχανισμούς για να ε, καμουφλάρουν την υποδύναμη. Εγώ αυτό κατάλαβα. Έχω την εντύπωση ότι η ισχύ ενό κινητήρα και αυτό το αναφέρει και η έκθεση, δεν είναι ένα ε, ε, στοιχείο ε, το οποίο καθορίζει τη δυνα... αληφτική δυνατότητα του σκάφους ή του τι πραγματικά αλλιεύει το σκάφος. Γιατί εφόσον υπάρχουν ποσοστώσεις συγκεκριμένες, είτε έχει μεγάλο κινητήρα είτε έχει μικρό το συγκεκριμένο σκάφος, δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό, την ποσόστοση που του έχει χορηγηθεί. Εντάξει, μπορεί να φτάσει νωρίτερα στο λιμάνι, μπορεί ίσως να ψαρέψει πιο γρήγορα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μία ποσόστοση έχει και αυτή είναι που ισχύει. αν είχαν περιορισμό στις ημέρες κατά τις οποίες μπορούν να αλλιεύουν, ναι, εκεί θα είχε επιρροή, γιατί θα μπορούσε να ε, ε, αλλιεύσει, ας πούμε, περισσότερο στη διάρκεια των ίδιων ημερών, αν είχε πιο ισχυρό κινητήρα, αλλά εκεί έχει, ίσως, αν έχουμε ένα μεικτό σύστημα με ποσοστώσεις και αλλιευτική προσπάθεια, πιστεύω πως θα έπρεπε ότι ένα καλύτερο κινητήρα δίνει περισσότερη ασφάλεια στον καπετάνιο και στο πλήρωμα. Γιατί αν κανείς πρέπει να ξεφύγει στην τρικυμία, ξεφεύγει πιο εύκολα με ένα δυνατό κινητήρα από ότι με έναν πιο αδύναμο δεν ξέρω αν αυτό δηλαδή έχει να κάνει με την υπεραλίευση και πρέπει να το συζητήσουμε και με το εκπροσώπους του τομέα. Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ε, περιπτώσεις, γιατί το φαινόμενο αυτό έχει λάβει τόσο ευρείες διαστάσεις. Δεν θέλω δηλαδή να προτρέξουμε ε, ε, και να φτάσουμε σε πορίσματα, γιατί κομμάτι της έκθεσης δεν το κατάλαβα, είναι πολύ περίπλοκο, αλλά και στην προοπτική των ε, κλιματικών αλλαγών για τις οποίες τόσο γίνεται λόγος ε, θα θέλαμε ίσως να έχουμε κινητήρες πιο αποτελεσματικούς από την άποψη των εκπομπών και, και αυτή την ευκαιρία για να πω ότι χρειάζεται να έχουμε πιο αποτελεσματικούς κινητήρες και όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας αλλά και όσον αφορά την χαμηλότερη ρήπανση. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Η Ρούς έχει το λόγο. Το Δεκέμβριο του 2018 το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν τα, τα ΤΑΚ. 90% των αλλιευμάτων δεν ανταποκρίνονται στους στόχους. Τώρα, εδώ, αυτό είναι, μια προβληματι... είναι ένα προβληματικό σημείο. Αυτά όλα συνέβησαν 8 μήνες πριν. Η Επιτροπή τώρα, με αυτήν την μελέτη, στο πρώτο σημείο βλέπουμε ότι 51% των σκαφών που εξετάστηκαν έχουν μεγαλύτερη ισχύ κινητήρα από ό,τι έχουν δηλώσει. Είναι τα, τα κράτη-μέλη της Μεσογείου που δείχνουν να μην συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Οι μετρήσεις που έγιναν δεν ήταν ακριβείς. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν, τόσο ώστε η επαλήθευση της μέτρησης του, της ισχύς του κινητήρα να είναι ακριβής και πώς αυτό βοηθάει στην υπερεκμετάλλευση των στόκ. Αν δεν είναι ακριβής η ισχύ του κινητήρα. Οι επιδοτήσεις από το Ταμείο πριν τις δώσουμε δεν θα πρέπει να εξετάσουμε τι είδους ισχύ χρησιμοποιείται πριν αποφασίσουμε να δώσουμε χρήματα για καινούριου κινητήρες, πριν αποφασίσουμε να δώσουμε επιδοτήσεις για αντικατάσταση κινητήρων στα σκάφη. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα πριν ζητήσω από την ε, Κομισιόν να απαντήσει. Ο κύριος Μιγιανμόν, κατά τη γνώμη μου, έχει γύρει κάποια σημαντικά ζητήματα και παρατήρησα επίσης ότι ένα από τα σημεία που θίγετε και εσείς στην έκθεσή σας είναι ότι πέρα από τις άλλες ατέλειες υπάρχει και μη συνοχή, μη συνέπεια μεταξύ της, της μέτρησης. Τι μετράμε, τη δυνατότητα σε μάκρος χρόνου να φτάνει μια συγκεκριμένη ταχύτητα ή μετράμε την επιτάχυνση, για παράδειγμα, σε μια δεδομένη στιγμή. Επομένως, υπάρχει και μια σάφια στο πώς θα γίνονται οι πιστοποιήσεις αυτές. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό ελέγχου, κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την νομοθεσία αυτή ή να καθίσουμε να περιμένουμε κι άλλες έρευνες Ωστόσο, στο συγκεκριμένο κανονισμό, μόλι περάσουμε το συγκεκριμένο κανονισμό ελέγχου, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε. Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει με δεδομένε τι δυσκολίε εδώ είναι ότι οι αληφτικέ προσπάθειε χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολύ καλό. Τι γίνεται με τα κράτη-μέλη που δεν χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό. Αυτό είναι ένας τρόπος για να εξασφαλίζουμε, για να προστατεύουμε τα στόκ και να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει βιώσιμη απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, υπενήσεστε ότι επιπλέον έλεγχοι θα γίνουν. Ίσως θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και με τη νέα επιτροπή που θα αναλάβει δράση. Μήπως θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για όλες τις ερωτήσεις ε, που έγιναν. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο σας διαβεβαιώ ότι τουλάχιστον στο δικό μας το επίπεδο αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα και παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά αυτήν την ε, μελέτη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Τώρα, για το θέμα του κυρίου Μιγιανμόν είναι σαφές ότι εντάξει, είναι τεχνικό το ζήτημα, το αναγνωρίζω και για μένα. Αλλά δεν πρέπει να είναι δικαιολογία για να μην ε, κάνουμε τίποτα. Όλοι αντιλαμβάνονται την σημασία αυτού του ζητήματος. Ε, πέρα από την υποδύναμη της μηχανής ε, και το να είναι μεγαλύτερη από την δηλωμένη στην άδεια. Και βεβαίως ε, ακόμα και πριν γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα προτείναμε μία αναθεώρηση του συστήματος ε, για να είναι λιγότερο επιβαραντικό για τις αρχές γιατί τώρα οι αρχές πρέπει να κάνουν κάποια σχέδια δειγματοληψίας και μετά φυσικούς ελέγχους. Γιατί βεβαίως αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται εξωτερικοί σύμβουλοι και εμείς καταλήξαμε στην πρόταση να υπάρχουν συσκευές που θα παρακολουθούν συνεχώς την υποδύναμη. Είναι λοιπόν σαφές ότι οι συσκευές αυτές έχουν ένα κόστος και για τον ίδιο ακριβώς λόγο έχουμε βάλει μία διάταξη στην ε, νέα πρόταση για μία παρέκκληση για την χρηματοδότηση του EMFF ε, που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχουν ε, τέτοιες διατάξεις για υποχρεωτικό ελεγχό. Γι' αυτό έχουμε εισαγαγεί μια παρέκκληση για την συνεχή παρακολούθηση της υποδύναμης έτσι ώστε αν αυτή μειωθεί στο μέλλον τα κράτη-μέλη θα έχουν την δυνατότητα να δώσουν επιχορηγήσεις ε, σε σκάφη που θα έχουν αυτές τις διατάξεις όπως έχει γίνει και με τη τηλεόραση κλειστού κυκλώματος. και βεβαίως υπάρχουν λασκάφιο που ίσω ίσως άλλοι τύποι ελέγχων και θα έπρεπε ακριβώς να δούμε την ε, μελέτη. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρατε κύριε Πρόεδρε στην αρχή της παρέμβασής σας ήταν ακριβώς τα αποτελέσματα και το ότι η μελέτη επισημαίνει την ε, πιθανή παραποίηση των δεδομένων του κατασκευαστή και από τις ε, εταιρείες πιστοποίησης. Ε, τότε δεν είχαμε βεβαίως βεβαίω τα αποτελέσματα της μελέτης, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης. Και μετά το θέμα για τις ποσοστώσεις ε, και τους ε, φορούς ε, που είναι θα έλεγα ο τρόπος με τον οποίο μετράμε την βιωσιμότητα των αποθεμάτων αλλά πρώτον όπως είπα υπάρχουν διάφορα καθεστώτα τα οποία ισχύουν και δεν θα πρέπει ακριβώς να τα ξεχνάμε σε διάφορους αλευτικούς ε, τομείς ε, στα ευρωπαϊκά ύδατα. Δεύτερον, για να είμαι ειλικρινής, ε, και αυτό είναι μια... αυτή είναι... Αυτός είναι ο λόγος της πρότασης. Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι για τα δεδομένα αυτά. Αν υπήρχε η βεβαιότητα ότι πραγματικά όλα τα αλλιεύματα καταγράφονται, τότε θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε ότι θα ξεφορτωθούμε κάποιους κανόνες που ούτως ή άλλως δεν είναι το αντικείμενο του κανονισμού, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για να έχουμε κάποια βεβαιότητα, για να υπάρχει πλήρης καταγραφή και για να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις βεβαίως, αν υπάρχει υπερβολική ισχύς, υπάρχει το κίνητρο να ψαρεύει κανείς περισσότερο και πιθανώς και να απορρίπτει αλλιεύματα. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί αυτό υπόψη. Συχνά επίσης ε, Ε, συμβαίνει το εξή. Ε, η ασφάλεια είναι γενής, δηλαδή το βασικό το σκάφος το οποίο χρησιμοποιείται ε, χρησιμοποιείται και για την ασφάλεια του πληρώματος, έτσι, στην περίπτωση που χαλάσει ο καιρός. Αλλά βεβαίως οι άλλες λειτουργίες εντός του σκάφους μπορεί να έχουν τις λεγόμενους βοηθητικούς κινητήρες και βεβαίως ε, αυτοί δεν συνυπολογίζονται στην υποδύναμη του κινητήρα και στα όρια τα συνολικά. Δηλαδή υπάρχει ο κύριος κινητήρας και η βοηθητική. Δεν συνυπολογίζονται όμως αυτοί στο όριο. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Για τις επιδοτήσεις δεν ξέρω αν η Ελίζα θέλει να πει κάτι για τον ορισμό της υποδυναμίας... Ε, ο πρόεδρος, να αναφερθώ, να ζητήσω μια διευκρίνηση. Γιατί αναφέρατε τις, ε, τους βοηθητικούς κινητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν ε, τον κύριο κινητήρα. Γιατί τις αναφέρετε αν δεν μετράνε. Ε, μπορεί να υπάρχουν αλλά δεν ε, συνεισφέρουν στην προώθηση του σκάφους και άρα στην αλληλεία Βελτιώνουν ε, τις συνθήκες υγιεινής, εργασίας ή την ποιότητα των προϊόντων. Ναι, για το θέμα των επιδοτήσεων και την παρέμβαση της κυρίας Χούς. Συμφωνώ πλήρως με αυτό το οποίο είπατε ότι έχουμε μια πρόταση στο σχετικό ταμείο για την ε, στήριξη επενδύσεων στην ασφάλεια, για την αντικατάσταση κινητήρων, ε, υπό όρους ε, βεβαίως. Υπάρχει μείωση της ισχύω του κινητήρα και υπάρχει και μια πραγματική επαλήθευση. Είναι απογοητευτικό το ότι οι διατάξεις αυτές πλέον δεν είναι στην συζήτηση με τους ε, συνομοθέτες. Πρέπει να δούμε πώς ε, θα εξελιχθεί ο τριμερής διάλογος, αλλά προφανώς εάν καταλήξουμε με ένα ταμείο στο οποίο μπορεί να αντικατασταθεί ο κινητήρας χωρίς μείωση της ισχύω και χωρίς ε, έλεγχο, επαλήθευση, όπως ανέφερε η συνάδελφος, θα Έχουμε λίγα πράγματα για να μπορέσουμε να πούμε στην περίπτωση στην οποία θα αυξηθεί η ε, δυνατότητα του στόλου. Και έρχομαι σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μιγιάν μόνο ότι πράγματι είναι υποκειμενικοί παράγοντες ε, το... η κόρη ενός ε, σκάφους και η υποδύναμη. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρούμε άλλους δείκτες τους οποίους θα αποδεχτούν και στους οποίους θα συνενέσουν ε, οι επιστήμονε οι ψαράδε κτλ. Το που χρησιμοποιούμε για την ώρα αυτού του δύο δείκτε για να μετρήσουμε την αλληλευτική ικανότητα. Αν λοιπόν το ένα, το οποίο είναι η επαλήθευση της ισχύω του κινητήρα δεν υπάρχει, δεν θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι δυνατότητε του στόλου. Και αυτό έχει σημασία. Ε, πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες του στόλου, γιατί οι ποσοστώσεις δεν είναι ο μόνος ο τρόπος, όπως αναφέρθηκε. Έχουμε πολλούς στόλους, πολλές λεκάνες που δεν ρυθμίζονται με ε, μέγιστα επιτρεπόμενα λεύματα και ποσοστώσεις και πρέπει ακριβώς να μπορούμε να αξιολογούμε ποιες είναι οι δυνατότητες του στόλου. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά βλέπετε τι ωραία περνάμε εδώ πέρα. Ε, ήρθε η Κομισιόν στην προηγούμενη παρουσίαση και σας είπε προχωράμε, πλησίστη προς την βιωσιμότητα και τώρα ήρθε εδώ πέρα και τα βάψε όλα μαύρα. Ελπίζω λοιπόν να δοθεί προτεραιότητα στο ζήτημα και να επανέλθουμε με κάποιες συστάσεις για το τι πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Item 10, which is the... Σημείο 10 σύναψη συμφωνίας ελευθερίου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και της Σοσιαλιστική Δημοκρατίας του Βιετνάμ. Θα γνωρίζετε ότι η Επιτροπή μας προετοιμάζει μια γνώμοδότηση για την σύναψη αυτής της συμφωνία, κύριο Μπατόλο των Σοσιαλδημοκρατών είναι ο εισηγητή και αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ πέρα είναι ότι ενώ έχει πολλά ωφέλη η εμπορική αυτή η συμφωνία, το Βιετνάμ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια διαδικασία κίτρινης κάρτας για μα, δηλωτή και παράνομη αλία. Και έχουμε πολύ σοβαρές επιφυλάξεις ε, για να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια συμφωνία μέχρι να, αναφερθεί, μέχρι να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο τώρα στον εκπρόσωπο εδώ πέρα, της Κομισιόν, τον κύριο Πίτερ Μπέτς. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας για το ενδιαφέρον. Έχουμε διαπραγματευτεί δύο τέτοιες ε, συμφωνίες. Η μία είναι και προστασίας ε, των επενδύσεων και οι δύο υπεγράψαν 30 Ιουνίου και αποτέλεσαν ορόσημο στις ε, σχέσεις μας. Όταν υπογράφηκαν αυτές οι συμφωνίες, το Βιετνάμ έβγαινε από την απομόνωση. Έκτοτε το Βιετνάμ ζει ριζική έναν ριζικό οικονομικό μετασχηματισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντικός εταίρος ε, του Βιετνάμ και τώρα έχουμε μία ευρύτατη συμφωνία που είναι αμοιβαίως υποφιλής ε, και απόδειξη γι' αυτό είναι η συμφωνία που τέθει ενισχύει τον Οκτώβριο του 2016. Η εμπορική συμφωνία θα ενισχύσει την συνεργασία μας και θα αποτελέσει έναν τρόπο για να ενισχύσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις. Οι συμφωνίες αυτές είναι οι πιο φιλόδοξες συμφωνίες που έχει συνάψει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι πολίτες θα ωφεληθούν από την πρόσβαση στην αγορά 100 εκατομμυρίων κατοίκων που αυξάνεται και αναπτύσσεται εντός του ΑΣΕΑΝ και έχει μια, ένα πάρα πολύ νεανικό και δυναμικό εργατικό δυναμικό. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο στοιχείο επαφής με την Νοτιοανατολική Ασία μετά τη συμφωνία με την Σιγκαπούρη. Βεβαίως ε, Δεδομένου του ότι υφίσταται και πίεση το πολυμερέ εμπορικό σύστημα, οι συμφωνίε αυτέ δείχνουν πω είμαστε προσιλωμένοι σε ένα ανοιχτό εμπόριο με κανόνε και μαζί με τη δυνατότητα να αυξηθεί το εμπόριο, να στηρίξουμε την ανάπτυξη και στι δύο πλευρές και θα ωφεληθούν ε, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και καταναλωτές. Ε, μιλάμε για πρόσβαση στις ε, αγορές αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων προμηθειών και κανόνες όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, διευκόνες τελωνίων και τεχνικά, εμπο, τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο. Έχουμε λάβει υπόψη και τις σχετικές ε, ευαισθησίες, παραδείγματο χάρη τον συσκευασμένο τόνο και το σουρίμι, τα οποία αποκλείονται από την πλήρη απελευθέρωση και θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιορισμένες ε, ποσοστώσεις. Άλλα είδη ψαριών ε, θα απελευθερωθούν μετά από τρία χρόνια μόνο και το Βιετνάμ με τη σειρά του θα καταργήσει σταδιακά τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αλληλευτικά προϊόντα. Έχουμε επίσης ένα κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης που στόχο έχει ακριβώς την προστασία της περιβάλλοντος ε, και τονίζει και την κλιματική αλλαγή και είναι εκπληκτικό το ότι για πρώτη φορά έχουμε ε, ένα τέτοιο κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη με μια αναπτυσσόμενη χώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και πλησιάζει τα κεφάλαια που έχουμε συνυπογράψει με χώρες όπως ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Με το κεφάλαιο αυτό, περί βιώσιμης ανάπτυξης, και οι δύο πλευρές δεσμεύονται για να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλασσίων πόρων και των προϊόντων ηχθειοκαλλιέργειας. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για συμμόρφωση με διεθνείς συμφωνίες και για συνεργασία εντός περιφερειακών οργανισμών αλληλείας. Επίσης το κεφάλαιο περιέχει κάποιες δεσμεύσεις που αφορούν την καταπολέμηση της λαθραλίας. το Βιετνάμ είχε επισημανθεί ως μη συνεργάσιμη χώρα στην καταπολέμηση της, αλίας, αλλά, της λαθραλίας, αλλά εν τω μεταξύ έχει επιδείξει μεγάλη διάθεση για συμμόρφωση. Έχει υπάρξει ένας νέος νόμος περί αλίες και εφαρμοστικός κανονισμός. Πρόκειται για ένα πρώτο και θεμελιώδες βήμα στην οικοδόμηση μιας νέας πολιτικής για να καταπολεμηθεί η λαθραλία στο Βιετνάμ όμως. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να υπάρξει εφαρμογή και έλεγχος των δραστηριοτήτων και των σκαφών που λειτουργούν στους ε, λιμένες ε, του Βιετνάμ. Η Επιτροπή Αλληλείας ε, της προηγούμενου κοινοβουλίου επισκέφθηκε το Βιετνάμ πέρσι τον Οκτώβριο και εξέφρασε την εκτίμησή της για τις προσπάθειες του Βιετνάμ για την καταπολέμηση της λαθραλίας και είπε ότι θα συνεχίσει να διεξάγει έναν επικοδομητικό διάλογο με τη χώρα. Τώρα η Κομισιόν θα συνεργαστεί στενά με τις αρχές του Βιετνάμ έτσι ώστε η χώρα να είναι πλήρω προετοιμασμένη για να εφαρμόσει αυτό το κεφάλαιο να δημιουργηθούν οι κατάλληλε διοικητικέ δομέ στο επίπεδο κράτου και κοινωνία των πολιτών Μόλι η συμφωνία αυτή τεθεί ενισχύει ελπίζουμε να συμφωνήσει γρήγορα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε οι επιχειρήσει ε, και οι καταναλωτέ να μπορούν να ωφεληθούν το συντομότερο δυνατόν και να συνεχίσουμε να έχουμε τι επαφές αυτές ε, που θα διατηρήσουν το Βιετνάμ σε μια πορεία μεταρρυθμίσεων. Κατόπιν ε, η συμφωνία αυτή θα πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενώ η Συμφωνία προστασία των Επενδύσεων πρώτα απ' όλα θα απαιτήσει την κύρωση από όλα τα κράτη-μέλη πριν ε, την συνάψει το Συμβούλιο. Πηγαίνοντα ε, προς ε, την κύρωση, έχουμε τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω επαφές με την χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Κότς. Επιβεβαιώνεται ότι η Κομισιόν εξακολουθεί να έχει μια διαδικασία κίτρινης κάρτας για την λαθραλία στο Βιετνάμ. Ναι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαρτελέ, ναι, ο εισηγητής μας, σωστά, σωστά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Η συμφωνία αυτή ελευθεροπορίου με το Βιετνάμ είναι μια ευκαιρία για τον ε, τομέα της αλληλείας στην Ήπειρό μας σίγουρα και για την εσωτερική μας αγορά. Ωστόσο, είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει όλο της το κύρος ε, και το βάρος της ως παγκόσμιος ε, παίκτης, ώστε να αποκομίσει οικονομικά ωφέλη από αυτή τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, αλλά και την προστασία του τομέα της αλληλείας, αλλά και των πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Θα πρέπει καταρχάς να θεωρήσουμε θετικό το γεγονός ότι η Συμφωνία αναγνωρίζει τη σημασία μιας βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσίων πόρων, καθώς όπως τονίστηκε τονίζεται μάλλον στο κεφάλαιο 13 σημείο 9. Θεωρώ κατά δεύτερο λόγο θετική τη δέσμευση των δύο μερών ώστε να αναχαιτιστεί η παράνομη ε, και μη ρυθμιζόμενη ελία. Είναι σίγουρα καλό νέο το αίτημα από πλευρά τη κυβέρνηση του Βιετνάμ να μπει ω μόνιμο μέλος της Επιτροπή Αλληλεία του Ειρηνικού του κέντρου ε, δυτικού ε, ειρηνικού. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο στενή συνεργασία ώστε να αναχαιτιστούν αποτελεσματικά αυτά τα φαινόμενα όπως ρητά αναφέρονται στην παράγραφο Β του δεύτερου σημείου του άρθρου 10.9. Ε, Τέλος, πάντοτε σε σχέση με την καταπολέμηση της παράνομη παράνομης είναι σίγουρα θετικές οι προσπάθειες της κυβέρνησης του Βιετνάμ ώστε να προσαρμόσει την εσωτερική της νομοθεσία η υιοθέτηση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τον ε, αλευτικό τομέα και για τη δημιουργία δομών ε, συντονισμού των προσπαθειών κατά πολέμηση παράνομη αλληλεία είναι ε, βήματα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν κάποια αρνητικά στοιχεία και κενά που πρέπει να καλυφθούν, όπω. το υπερβολικό μέγεθος του στόλου ή η υπερβολική εκμετάλλευση των ε, αλληλευτικών πόρων. Προς προς αυτό, τα μέτρα που προτείνονται όπω η κίτρινη κάρτα, που προτάθηκε το 2017 θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένους στόχους και οδικούς χάρτες για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Επίσης, οι προτιμησιακές ε, ε τιμές που προσφέρονται μέσω της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών να δίνονται αλλά με αντίτιμο συγκεκριμένα μέτρα και με μέρημνα ώστε να μειωθεί ο ελευτικός στόλος της χώρας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να ασκεί διαρκή πίεση ώστε οι αρχές του Βιετνάμ να, να, να παρακολουθούν εκ του σύνοικης την πορεία του στόλου τους και να εξασφαλίζουν την ανεχνευσιμότητα των προϊόντων που, προορίζονται για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό το να εξασφαλίσουμε εγγυήσει, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα αναστολής προσωρινής της συμφωνίας στην περίπτωση που η Βιετναμέζικη πλευρά δεν ανταποκρίνεται στους όρους βιώσιμη βιώσιμης ανάπτυξης που έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εισηγητής λοιπόν για αυτή τη γνωμοδότηση, στο κείμενό μου θα κινηθώ με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές που μόλις σας ανέφερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι να μπορέσω ε, να συνεργαστώ επικοδομητικά μαζί σας με βάση τις τροπολογίες που θα υποβάλλετε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Μπάρτολο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία αυτή μας δίνει πολλές ευκαιρίες στον τομέα του εμπορίου και οπωσδήποτε 99% των δασμών θα εξαφανιστούν και θα έχουμε ανάπτυξη και στις δύο πλευρές και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θα έχουμε λοιπόν ίσους όρους ανταγωνισμού στον τομέα της υγιεινής, ε, της ασφάλειας των τροφίμων και των κοινωνικών ζητημάτων. Βεβαίως, ε, από πλευρά της Επιτροπής μας έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το πρόβλημα που υπάρχει με την λαθραλία στο Βιετνάμ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις ε, διαδικασίες αυτές ε, και δεύτερον να έχουμε ξεχωριστές διαδικασίες για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να παραμείνουν διαχωρισμένες. Η συμφωνία αυτή ελευθερου εμπορίου μας προσφέρει πολλές ευκαιρίες όχι μόνο για τον τομέα της αλίας αλλά και για τους άλλους κλάδους και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Μόλις το είπα άλλωστε. Και αντιλαμβάνομαι ότι η διαδικασία στο πλαίσιο του IO πηγαίνει και εξελίσσεται όμαλα αλλά θα πρέπει να συμπληρωθεί με την σχετική νομοθεσία η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί με παρακολούθηση και μέτρα ελέγχου. Οπότε θα πρέπει να είμαστε κάπως ε, επιφυλακτικοί και αντιλαμβάνομαι από την ε, Digimare πως θα είναι σε συνεχή επαφή με το Βιετνάμ. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία και αναμένω την επόμενη έκθεση σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ήδη έχετε καταλάβει ότι έχω φρικτή προφορά. Ε, εμένα λέτε, ναι κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε το ονοματάκι σας για να τα ακούσω. Ε, bien. Muchísimas gracias, Presidente. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. μάλιστα. Ε, θετικά εκτιμούμε αυτή την ε, συμφωνία ελεύθερο εμπορίο, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής μας υπάρχει ε, μια κίτρινη κάρτα και αυτό μας προκαλεί ανησυχίες. Ε, η Κομισιόν μας ενημέρωσε ότι για το γεγονό γεγονός ότι το Βιετνάμ έχει κάνει προόδο. Υπήρξε και μια πρόσφατη αποστολή του Κοινοβουλίου για να δούμε επιτόπου τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την δημιουργία θεσμικών δομών ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτή την νομοθεσία για την οποία μιλήσαμε. Όμως υπάρχει κάτι που μας ανησυχεί σε αυτή την Επιτροπή και είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ήδη έχουμε βρεθεί όσον αφορά την εφαρμογή της ε, συμφωνίας και εξακολουθεί να μην υπάρχει επαρκής έλεγχος. Τώρα το θέμα της βιωσιμότητας που αναφέρθηκε. Υπάρχει έλλειψη διαχείρισης ε, του αλληλευτικής ε, προσπάθειας και αυτό προκαλεί την ανησυχία μας όσον αφορά την αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στη δική μας ε, αλληλευτική βιομηχανία που οφείλει να τηρεί τους, τις ε, ευρωπαϊκές νομοθεσίες, αλλά και κυρίως γιατί ε, ανησυχούν οι Ευρωπαίοι πολίτες που ανησυχούν για την βιώσιμη προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουν. Στην αποστολή του Νοεμβρίου της Επιτροπής μας, ποια είναι τα στοιχεία και τα κριτήρια ε, και οι ενέργειες που έγιναν ώστε να μπορέσουμε παρκώς να επαληθεύσουμε τις προόδους που έχουν γίνει στο σύστημα ελέγχου και ποιες είναι οι εγγυήσει ότι το ελεύθερο εμπόριο άλλων προϊόντων δεν ε, ε, θα παρεμποδιστεί από την ανάγκη, για παράδειγμα, απαγόρευσης εισαγωγής κάποιων προϊόντων από το Βιετνάμ. Να δούμε δηλαδή αν υπάρχει ρήτρα ε, αναστολής της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλές ε, και συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κύριε Σάλιβαν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Για να συνεχίσω ε, σε σχέση με, τον ε, πράσινη, ε, με την κίτρινη κάρτα που είναι ένα σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν μίλησε για μια ανοιχτή υπόθεση και για έναν ε, εμπορικό μηχανισμό που βασίζεται σε κανόνε. Αλλά όπω είπε και ο συνάδελφο, όσον αφορά τον ανταγωνισμό, πώ μπορεί να είναι δίκαιο εάν οι Βιετναμέζοι έχουν ένα σύστημα με κίτρινη κάρτα, το οποίο ε, στην ουσία ε, θέτει σε μειονεκτική θέση το δικό μας σύστημα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έπειτα λένε ότι βασίζεται το σύστημά τους σε κανόνες. Θα ήθελα να ξέρω από την Κομισιόν τι κάνουν ώστε να εξασφαλίσουν ότι μια αναπτυσσόμενη, γρήγορα αναπτυσσόμενη χώρα από οικονομικής άποψης πώς θα εξασφαλίσει η Κομισιόν ότι θα υπάρχει όντως ένα, θα επικρατήσει μάλλον ένα δίκαιο σύστημα που βασίζεται σε κανόνες για μια χώρα όπως το Βιετνάμ. Μάλιστα, δεν βλέπω κανέναν άλλο να ζητά το λόγο. Κύριε Κότς, λοιπόν, εσείς μας παρουσιάσατε μία ε, ισχυρά επιχειρήματα με βάση τα οποία θα πρέπει να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία, αλλά είπατε ότι υπάρχει πρόοδος ε, όσον αφορά την καταπολάμηση του IUU, της παράνομης και ε, ανεξέλεγκτης αλληλείας, όμως υπάρχουν διάφορες ομάδες που εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις και φαντάζομαι ότι αυτό δεν, είναι, και δεν σας εκπλήσει γιατί τώρα θα πρέπει οι διαπραγματευτές ε, της Ένωσης ε, να έχουν το πάνω χέρι στο να αλλάξουν τις πολιτικές της χώρας αυτής προς το καλύτερο. Μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, βεβαίως. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπα, η συμφωνία που θα είναι η τέταρτη που θα έχουμε συνάψει με μια ασιατική χώρα μετά από την Κορέα, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη είναι οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας αλλά και πολιτικής σημασίας και αυτό όχι μόνο στον τομέα της παράνομης ανεξέλεγκτης αλληλείας αλλά και για τα εργατικά δικαιώματα το βλέπουμε στο πολιτικό τομέα, το βλέπουμε για το κλίμα. Το Βιετνάμ ε, υπέγραψε την Συμφωνία του Παρισιού, πράγμα που δεν ξέρουμε αν θα ήταν δυνατόν ε, αν δεν είχε υπάρξει αυτή η συμφωνία βλέπουμε την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας ως γενικό στόχο όχι μόνο στην Ένωση αλλά και διεθνώς και στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ έχει κάνει αξιόπιστες προσπάθειες, δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα, γι' αυτό και τους δώσαμε κίτρινη κάρτα. Είναι μια διαδικασία αλλά όπως ε, είπε και ένας βουλευτής, είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Από τη μια πλευρά έχουμε βεβαίως ε, την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και από την άλλη έχουμε και τη διαδικασία της καταπολέμησης ε, της παράνομης αλίας. Οι δυο προχωρούν παράλληλα. Η εμπορική συμφωνία μας δείχνει ισχυρή δέσμευση για, από πλευρά Βιετνάμ να συνεργαστεί για την καταπολέμηση παράνομη αλληλεία και να τηρήσει τι υποχρεώσει του ε, με βάση τι διεθνεί συμβάσει. Και ε, αναφέρουμε στην συνάδελφο τη DG Mare, αν είναι έτοιμη για να συμπληρώσει στις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως έλεγε και ο Πίτερ, πρέπει πραγματικά να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο προγράμματα. Από τη μία έχουμε την επικύρωση και την εφαρμογή της ελεύθερης συμφωνίας συναλλογών και από την άλλη έχουμε τους διαλόγους στα πλαίσια της διαδικασίας παράνομης λαθραλίας. Α, μόλις θεσπιστεί μια κίτρινη κάρτα, μόλις υιοθετηθεί μια κίτρινη κάρτα με μια τρίτη χώρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξεκινάει ένας επίσημος διάλογος. Και με το διάλογο αυτό ο διάλογος αυτός μάλλον συνοδεύεται και από ένα σχέδιο δράσης και η δέσμευσή μας μέσω της επεξεργασίας αυτής είναι να παρακολουθήσουμε από κοντά τι ακριβώς κάνει το Βιετνάμ σε σχέση με αυτό το σχέδιο δράσης που ορίζουμε. Η εκπλήρωση των κανόνων για την παράνομη λαθραλία είναι τελείως ανεξάρτητη από τους, τις δεσμεύσεις που ορίζει η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, το FTA. Υπό την έννοια ότι αν έχουμε μια κίτρινη κάρτα, αν θα παραμείνει όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο από τη Συμφωνία Εμπορίου που θα υπογράψουμε. Και αυτό είναι που θέλω να ξεκαθαρίσω. Οι κανόνες για τη λαθραλία. Κάθε αλληλευτικό προϊόν που εξάγεται θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ότι δεν προέρχεται από παράνομη λαθραλία. Το ίδιο ισχύει και για τι υγειονομικέ συνθήκε των εισαγωγών που κάνουμε. Υπάρχει μια σειρά από κανόνε που θα πρέπει να πληρούνται, ούτω ώστε να μπορεί μια χώρα να εξάγει προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ανεξάρτητο από την συμφωνία. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονό ότι είναι μια διαδικασία και η Κομισιόν παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, ε, τις πρόοδους που σημειώνει το Βιετνάμ. Έχουν τροποποιήσει εντελώς ε, το νομικό πλαίσιο στο Βιετνάμ και τώρα είναι η στιγμή να ξεκινήσουν να το εφαρμόζουν, να ξεκινήσουν να το επιβάλλουν. Έχουμε ήδη δει κάποια θετικά βήματα, κάποιες θετικές εξελίξεις και είναι μίλουσα σημασίας αυτή τη στιγμή η έρευνα που θα κάνουμε τον Νοέμβριο. Εκεί θα δούμε σε πραγματικό χρόνο επιτόπου τι ακριβώς έχει γίνει και αυτό θα, θα σηματοδοτήσει και το μέλλον αυτής της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βιετνάμ σε σχέση με την ελαφραλία. Αυτό που ζητάμε από το Βιετνάμ είναι να μας δώσει αποτελέσματα, απτά αποτελέσματα σε κάθε σημείο του σχεδίου δράσης. Αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο σχέδιο δράσης της, ε, της ε, Κομισιόν. Α, σημειώνονται όλα αυτά τα σημεία και το γεγονός ότι το Βιετνάμ έχει σηματοδοτηθεί ως μη ε, συμμορφούμενη χώρα. Βεβαίω θα σας δώσουμε κάποιο feedback μόλις επιστρέψουμε από την αποστολή μας στο Βιετνάμ. Και πάλι όμως, εμείς υπογραμμίζουμε ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τη λαθραλία ανεξάρτητα από την ε, Συμφωνία Εμπορίου. Ευχαριστούμε. Επομένως υπάρχουν και κάποιες θετικές εξελίξεις. Ξέρουμε ότι το Βιετνάμ θέλει τη συμφωνία αυτή, όπως και εμείς άλλωστε. Αλλά το μήνυμα που θα πρέπει να σας δώσουμε εμείς και εσείς με τη σειρά σας στις αρχές του Βιετνάμ είναι ότι θέλουμε να πάψει η λαθραλία. Και θέλουμε οι κανόνες που αυτή τη στιγμή ορίζουν να εφαρμοστούν. Διαφορετικά δεν μπορούμε και εμείς να αγγιηθούμε την επικύρωση της συμφωνίας αυτής. Θα το συζητήσουμε και πάλι στις 2 Οκτωβρίου όταν ο κύριος Μπαρτόλο θα παρουσιάσει την εισήγησή του και στις 12 Δεκεμβρίου θα έχουμε ένα ψήφισμα, ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ελπίζω να μπορέσετε να μεταφέρετε το πνεύμα εδώ της Επιτροπής μας στις αρχές στο Βιετνάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Uh, Συνάδελφοι, σημείο 11 τώρα. Τρεις πράξεις κατεξουσιοδότηση υπό εξέταση. Το πρώτο έχει να κάνει με τη Σύμβαση Μελλοντικής Πολυμερούς Συνεργασίας στον τομέα της Αλίας στο Βόρειο-Ανατολικό Ατλαντικό. Ζητήσαμε δύο μήνες επιπλέον ε, περιθώριο εξέτασης για να δούμε κατά πόσο θα καταγραφούν ενστάσεις. Δεύτερο, Κομισιόν Η δεύτερη κατεξουσιοδότηση πράξη έχει να κάνει με την απόρριψη των αμοιβάδων και η τρίτη με τα βαθύβια αλληλευτικά προϊόντα. Έχουμε και άλλες τρεις πράξεις από την Κομισιόν που και πάλι συνδέονται με την απόρριψη, με τα σχέδια απόρριψης για βαθύβια αλληλευτικά προϊόντα στη Βόρεια Θάλασσα και στην ε, βορειοδυτική, στα βορειοδυτικά και στα νότιοδυτικά ύδατα. Να δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν τώρα. Ο κύριος Λουί Μαλέντο είναι. Όχι. Συγγνώμη. Διαφορετική σειρά των ομιλητών. Οκ, okay, ξεκινάμε με τον κανονισμό στην Μεσόγειο. Η κυρία Βαλερή Λέν έχει το λόγο. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα. Χαίρετε, χαίρομαι πολύ εκ μέρους της Κομισιόν να σας κάνω αυτήν την ε, παρουσίαση σήμερα για τις πράξεις κάτω εξουσιοδότησης. Πρώτα απ' όλα για το σχέδιο απόρριψης στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας και στο δεύτερο για τα βαθύβια είδη στο σύνολο της Μεσογείου. Ε, πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τα σχέδια απόρριψης, ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2019. Βρίσκεται στον πίνακα 3 των τεχνικών μέτρων για την Μεσόγειο. Γνωρίζετε ήδη ότι η κοινή πολιτική α, της Αλίας ορίζει ότι ο κανονισμός αυτός, το σχέδιο αυτό απόρριψης ισχύει τόσο για τους ψαράδες όσο και για τους ελέγχους. Αυτό το σχέδιο απόρριψης επιτρέπει ε, να λαμβάνονται υπόψη κάποιες ε, περιπτώσεις όπου υπάρχουν ε, παρακάμψεις, όταν υπάρχουν μίνιμουμ περιορισμών Σήμερα λοιπόν θέλω να σας παρουσιάσω τα στοιχεία που αφορούν την, ε, μεθο... την Μεσόγειο και συγκεκριμένα τα βαθύβια είδη. Είναι μια πράξη κάτω εξουσιοδότηση που προβλέπει την ε, επέκταση των ε, παρεκκλήσεων που υιοθετήσαμε πέρσι. Πέρσι υιοθετήσαμε κάποιες τέτοιου τύπου παρακάμψεις με επιστημονική συμβουλή πάντα σε επιστημονική βάση σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα είδη στόκ, πιο συγκεκριμένα... κάποια συγκεκριμένα είδη και οι παρακλήσεις μας βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες. Η Κομισιόν ήταν πολύ αυστηρή πάνω στον τομέα αυτό Ζητώντα να γίνουν επιστημονικές έρευνες από τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να μπορέσουν να επιδείξουν ε, συμμόρφωση με όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα. Λάβαμε λοιπόν μια σειρά από συστάσεις, τρεις συστάσεις από, τις, ε, από κάποιους περιφερειακούς οργανισμούς για τη διαχείριση της αλίας, πάντοτε από μεσογειακές χώρες, που υπέβαλαν ε, κάποιες, κάποια ερωτήματα σε σχέση με την επιβιωσιμότητα και τα ερωτήματα αυτά εξετάστηκαν με τρόπο ενδελεχή και αυτό που διαπιστώσαμε, αυτό που Αναρωτηθήκαμε είναι κατά πόσο αυτά τα είδη μπορούν να επιβιώσουν σε περίπτωση απόρριψης στη θάλασσα. Ένα άλλο θέμα που λάβαμε υπόψη μας ήταν η ανανέωση των παρακάψεων που αφορά τις εξαιρεσει. Κυρίω κυρίως ό,τι αφορά το μη εφικτό κόστος. Στην Μεσόγειο αντιμετωπίζουμε κάτι το οποίο αφορά τη Μεσόγειο. Συγκεκριμένα έχουμε μικρά σκάφη που μπορούν να φέρουν μικρό όγκο αλίας και υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να υπογνωμίσουμε είναι ότι στην Μεσόγειο δεν έχουμε τάκ. Επομένως, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο εφαρμόζεται στον Ατλαντικό, για παράδειγμα. Να λάβουμε δηλαδή υπόψη μας τα τάκ αυτά για τις απορρίψεις. Αυτό που ζήτησαμε από τα κράτη-μέλη λοιπόν ήταν να συνθέσουν κάποια στοιχεία για να μπορούν να στηρίξουν α, αυτήν την διαδικασία, αυτά τα σχέδια απόρριψης. Και έχουμε στα, στα χέρια μας αυτά τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να πούμε ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα πάνω στα πλοία σε αυτά τα μικρά πλοία, με αυτή την ιδιαιτερότητα της Μεσογείου που σας περιέγραψα, με ε, αποτέλεσμα να υπάρχει απόρριψη μικρών ποσοτήτων. Α, όλα αυτά επέτρεψαν στην ε, Κομισιόν να δώσει μια θετική γνώμη για αυτές τις παρακάμψεις για α, συγκεκριμένες ομάδες μεσογειακών κρατών. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι εδώ υπάρχει αρκετή επιστημονική βάση, εμπεριστατωμένη επιστημονική βάση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτά τα σχέδια απόρριψης, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις εξαιρέσεις, αυτές τις παρακάμψεις για τα βαθύβια είδη. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν εδώ είναι να παρατείνουμε αυτό που έχουμε ήδη οθετήσει. Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε τον κανονισμό αυτό πριν το τέλος του χρόνου. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει την υποχρέωση εκφόρτωσης ε, σε επίπεδο αρχών. Πρέπει να υιοθετήσουμε αυτή την πράξη εξουσιοδότηση για να μπορούμε να έχουμε έναν αποτελεσματικό έλεγχο τους πρώτους μήνες του ε, ερχόμενου χρόνου για να μπορέσει να εφαρμοστεί και η υποχρέωση εκφόρτωση. Σε ό,τι αφορά την άλλη ε, κατεξοδότηση πράξη πρόκειται για το σχέδιο για, τις, ε, για τα κηδόνια στα Ιταλικά ύδατα. Πρόκειται για ένα σχέδιο απόρριψης ε, το οποίο ε, ισχύει ε, θα ισχύει για τρία χρόνια και σκοπεύει να εξασφαλίσει την επιβίωση των αρχιβάδων αυτών στα Ιταλικά ύδατα αλλά και το μήνυμο μέγεθος από τα 25 εκατοστά στα 22 εκατοστά. Αυτή η πρόταση έγινε μέσω μιας κοινή σύστασης που συνέταξε η Ιταλική κυβέρνηση για τα Ιταλικά χωρικά ύδατα και αποκλειστικά τα ιταλικά χωρικά ύδατα και άρα η πρόταση αυτή βασίστηκε σε αποτελέσματα της εφαρμογής του προηγούμενου σχεδίου ε, πόρυψης και έτσι ε, επίσης κάποια μέτρα διατήρησης, συντήρησης μάλλον, τα οποία έχουν προταθεί από την Ιταλική κυβέρνηση, καθώς και ε, επιστημονικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί σε σχέση με την βιωσιμότητα. Ε, το ΣΤΕΦ, το επιστημονικό, η επιστημονική ομάδα, εξέτασε αυτή την πρόταση και κατέληξε στο ότι τα μέτρα που υιοθετήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου, βάση το προηγούμενο σχέδιο, επέτρεψαν την ανάπλαση του στόκ η Ιταλική κυβέρνηση μείωσε τον αριθμό των σκαφών, μείωσε την πίεση επί αυτού του αποθέματος διότι θέσπισε ένα σύστημα ε, ε, ε, ε, ποσόστοσης για κάθε σκάφος με περιορισμό του, ε, του αλλιεύματος από 600 κιλά σε 400 κιλά ανά ε, σκάφος. Σχέφηξαν ένα σύστημα VMS για τον εντοπισμό των σκαφών, ένα σύστημα ρήψης των αχιβάδων που ήταν μικρότερες από το επιτρεπόμενο μέγεθος, καθώς και επίσης ένα σύστημα ελέγχου στην εκφόρτωση. Το σύνολο λοιπόν αυτών των μέτρων επέτρεψε στο Επιστημονικό Συμβούλιο να διαπιστώσει ότι ο αντίκτυπος αυτού του συστήματος απόρριψης δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στο αποθεματικό αυτό και άρα στο αλίευμα αυτό και άρα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με αυτό το σχέδιο απόρριψης. Όσον αφορά την βιωσιμότητα, η Ιταλική κυβέρνηση υπέβαλε επιστημονικές μελέτες οι οποίες μας επέτρεψαν να ε, δηλώσουμε ότι η βιωσιμότητα αυτού του αποθέματος ε, είναι βέβαιη και ότι όταν ξαναπέσει στην θάλασσα ε, το κηδόνι μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του, ε, το κύκλο της ζωής του χωρίς πρόβλημα. Όσον αφορά το μήνυμο μέγεθος, επίσης το Επιστημονικό ε, Συμβούλιο θέσπισε ότι η μείωση του ελάχιστου μεγέθους δεν είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπλαση του αποθέματος και άρα μπορούσε να επιτραπεί η μείωση. Το σύνολο λοιπόν αυτών των στοιχείων, είτε πρόκειται για κοινωνικο-οικονομικά, είτε πρόκειται για επιστημονικά στοιχεία, επέτρεψαν στην Επιτροπή να προτείνει τη δημιουργία αυτού του σχεδίου απόρριψης για ένα χρόνο. Γιατί, ε, μόνο ένας χρόνος, γιατί ακριβώς θέλουμε οι επιστημονικές μελέτες να συνεχίσουν να γίνονται για να στοιχειοθετείται αυτή η εξαίρεση και στην επόμενη αίτηση εξαίρεσης να γίνει σύμφωνα με τον νέο κανονισμό με τα τεχνικά μέτρα που άρχισε να ισχύει στις 14 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Σας προτείνουμε λοιπόν να εγκρίνετε αυτό το σχέδιο ε, απόρριψης τόσο για την εξαίρεση όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος όσο και την διάρκεια του ενός έτους. Αυτές είναι οι δύο κατεξοδότησε πράξεις λοιπόν πρόεδρε που είναι πολύ σημαντικές. στο σχέδιο το απόρριψης για τα κυδόνια αφορά 500 σκάφη, ενώ η απόρριψη των βενθοπελαγικών ειδών αφορά χιλιάδες σκάφη σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Υπάρχουν ένα σωρό λοιπόν φορείς που θα ε, εφαρμόσουν αυτά τα συστήματα ε, και από οικονομικής και από νομικής άποψης θα πρέπει αυτά τα σχέδια απόρριψης να υιοθετηθούν όσο γίνεται πιο σύντομα, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν υποχρεώσεις εκφόρτωσης από την 1η Πρώτου Ευχαριστώ. Thank you. Any comment... Ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια από τα κράτη-μέλη. Η κυρία Κόντε, ευχαριστώ. Παραθέτω. Όσον αφορά τις χιβάδες, η οθότηση ε, του σχεδίου απόρριψης το 2016 έδωσε ωφέλη και στο οικονομικό και στο περιβαλλοντικό επίπεδο. Η μείωση των ημερησίων ορών ε, αλλιευσής ε, οδήγησε σε εξοικονομήσεις στα καύσιμα και επέτρεψε την καλύτερη εκμετάλλευση των αλλιευτικών ζωνών. Η Τεχνική Οικονομική Επιτροπή Αλλιείας διαπίστωσε ότι αυτό το καθεστώς εφαρμόζεται στα κηδόνια, ακόμα και αν μειωθεί το 20, από 25 εκατοστά στα 22 εκατοστά ε, παραμένει πάνω από το μέγεθος της πρώτης ορίμανσης ε, και άρα επιτρέπει την ανάπλαση του αποθέματος. Θεωρούμε Θεωρούμε λοιπόν λογική λογικό το αίτημα εξαίρεσης από το μήνυμο μέγεθος όσον αφορά την δυνατότητα ε, ε, της διατήρησης του στόκ ε, και ε, ε, επιτρέπεται για ένα χρόνο η μείωση του ελάχιστου μεγέθους των ε, αχιβάδων αυτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις εταιρείες μας, κυρίως για τη Βόρεια Αδριατική. Θα είχαμε προτιμήσει παράταση της εξαίρεσης για άλλα τρία χρόνια ή έστω για δύο. Είμαστε λοιπόν ε, ε, πέρ της καταξιδιώτησης πράξης και θέλω να καθησυχάσω τους Ισπανούς συναδέλφους ότι για την παράταση της εξαίρεσης ενός ή δύο ετών αυτή ε, εξυπηρετεί τη βελτίωση της ανάγνωσης των στοιχείων και ούτως ή άλλως ε, το κείμενο της κατεξουσιδότησης συμπράξης είναι, σωστό, είναι καλό έτσι και δεν χρειάζεται να δοθούν και άλλοι μήνες για την μελέτη. Δεν έχει δεν γίνει καμιά αναφορά στις προβληματικές της αγοράς γιατί η κατεξουσιδότηση συμπράξη προκύπτει από τον βασικό κανονισμό που δεν ασχολείται με αυτές τις πτυχές αλλά μόνο με τη ασχολείται μόνο με την προστασία του περιβάλλοντος και όχι με εμπορικά ζητήματα. Και άρα δεν θα ήθελα να καθυστερήσει η έγκριση αυτών των πράξεων μόνο και μόνο λόγω ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Um, uh, η κυρία Αγγιλέρα, ναι. Μόλις ακούσαμε μια παρουσίαση από πλευρά της, ε, κυρία, ε, της Κομισιόν για δύο από αυτές τις κατοεξιδότητες πράξεις και αυτής για τα βενθοπελογικά είδη. Άκουσα από κάποια μέλη ότι ανησυχούν ε, αυτή η πρόταση είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλο εύρος πεδίο εφαρμογή και ότι υπάρχει και ότι υπονοεί εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωση. Έχετε εσεί ερωτήσει για την Κομισιόν. Sí, Καταρχά, να ζητήσω συγγνώμη γιατί σήμερα ταυτόχρονα συνεδριάζει η Επιτροπή Γεωργίας, η Επιτροπή Αλίας και η Επιτροπή Αναφορών, όπου έπρεπε και εκεί να ε, παρέμβω. Δεν ήταν εύκολη η ατζέντα μου σήμερα. Ζητώ συγγνώμη, όμως με ενδιαφέρει πολύ αυτή η κατεξουσιοδότηση πράξη, ιδιαίτερα για τα ε, εισαχιβάδες και για την παράταση ενός έτους. Δεν μπόρεσα να ακούσω την Κομισιόν και δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση ε, χωρίς λόγο γιατί θέλω να διευκρινίσω το εξή. Εγώ προέρχομαι από την Ανδαλουσία και ήμουν και μέλος της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας ε, ε, όπου ε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον κόλπο του Κάντι. έχει σταματήσει η αλίευση της χιβάδας. Γιατί, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σωστό μέγεθος και αυτό με βάση επιστημονική μελέτη για έξι μήνες. Δηλαδή, ελήφθη αυτό το μέτρο για τον κόλπο του κάτι, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει αυτό το αλίευμα. Όπως είπα, κυρίως όσον αφορά το μέγεθος, αλλά και ε, για μία πιθανή υπεραλίευση. Ε, ε, και τώρα πάλι η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας πρέπει να λάβει μέτρα για τον κόλπο του Κάντιθ. Τι συμβαίνει τώρα, το να έχουμε το ίδιο προϊόν στην αγορά, γιατί η χιβάδα αυτή είναι πολύ μικρή ε, χιβάδα του κόλπου του Κάντιθ ή της Άρα λοιπόν μιλάμε για τον ίδιο αγορά. Η κατάσταση της αλληλείας στον κόλπο της Κάντιθ μου έλεγαν εμένα τότε εδώ και χρόνια όταν ήμουν μέλος της κυβέρνησης δεν καταλαβαίνουμε γιατί να ισχύει αυτό εδώ στον κόλπο του Κάντιθ ενώ στην Ιταλία υπάρχει αυτή η εξαίρεση και δεν χρειάζεται να τηρήσουν την υποχρέωση ε, μεγέθους. Ενώ όλοι ανταγωνιζόμαστε στην ίδια ευρωπαϊκή αγορά. Ήδη το έχω πει με την κυρία Κόντε. Έχω καταλάβει το επιχείρημά τη και τη είπα σήμερα το πρωί ότι θέλω να δω λεπτομέρειε την ε, περίοδο εφαρμογή και την ίδια την ε, κατεξουδότηση πράξη. Αλλά ότι θα ήθελα να ε, καταλάβουμε ότι αυτή η κατάσταση που διατηρείται εδώ και κάποια χρόνια και που επαναλαμβάνεται και πάλι δίνεται μια ακόμα παράταση για ένα χρόνο, δημιουργεί καταστάσεις επίμαχες με μια άλλη ζώνη ευρωπαϊκή που είναι ο κόλπος του Κάντιθ. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Δαλουσίας ε, έχει επιβάλει ένα σχέδιο ανάκτησης του αποθέματος. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να εξηγήσουμε τι συμβαίνει στον κόσμο εκεί. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να δοθεί αυτό το μέτρο το πρότεινε η Ιταλική κυβέρνηση, θα έχει τα επιχειρήματά της, δεν αφιβάλλω. Εγώ όμως θέλω να έχω τα απαραίτητα επιχειρήματα και εξηγήσει ώστε να πάω στον κόλπο του Κάντεθ και να τους πω, κοιτάξτε, το, ε, ε, ε, εκεί είναι 21 και εδώ είναι 25 και εδώ έχουμε να κάνουμε με την ίδια αγορά. Λοιπόν, θέλω να έχω εξηγήσει που να μπορούν να σταθούν και να τους τις δώσω. Εάν δεν καταλάβω και αν δεν έχω τέτοια επιχειρήματα στη διάθεσή μου, τότε θα χρειαστεί να καταψηφίσω. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί κάτι διαφορετικό σε μια ζώνη που ανταγωνίζεται στην ίδια ε, αγορά, την ευρωπαϊκή. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ποια είναι η διαφορετική κατάσταση για το ίδιο προϊόν. Όχ, όχ. Συναρπαστική συζήτηση. Κύριε Μελάτσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ άκουσα με πολύ προσοχή την εκπρόσωπο τη Επιτροπή που επιχειρηματολόγησε με στοιχεία. Αδιαφυσβήτητα και πιστεύω πως η αγορά, ο ανταγωνισμός, για να πω αυτές τις δύο λέξεις, δεν μπορεί να καθορίζεται από αυτήν εδώ την Επιτροπή. Και αυτό γιατί ο πρόσωπος της Επιτροπής μας διαβεβαίωσε, μάλλον πιστοποίησε με επιστημονικό τρόπο, ότι τα 22 το 22, αυτό το μαγικό νούμερο, επιτρέπει την αναπαραγωγή του στόκ των αχιβάδων αυτών. Δεν αλλάζει ε, καθόλου η κατάσταση και μάλιστα ε, παληθεύθηκε ότι η Ιταλική κυβέρνηση έλαβε τέτοια μέτρα ώστε να καταστεί συμβατή ε, αυτού του είδους η αλληλεία πιστεύω και γι' αυτό παρεμβαίνω. Δεν θέλω να ασκήσω υπεράσπιση και φτάνω στη δική μου πρόταση. Θεωρώ δεδομένο ότι εφόσον ακούσαμε αυτά τα στοιχεία δεν μπορούμε να το στείλουμε στο σπίτι του το θέμα, ενώ εφο... Ε, ε, επιστημονικά ε, αποδεικνύεται πως είναι κάτι το εφικτό. Εφόσον στατιστικά και επιστημονικά αποδεικνύεται πως μπορεί να γίνει, θα πρέπει να γίνει. Απλώ θα ήθελα να κάνω έκκληση στην Κομισιόν για τις δύο παραμέτρους. Η μία, η μία εξαίρεση δίρκεσε τρία χρόνια. Σήμερα προτείνει ακόμα ένα έτο εξαίρεση. Αλλά για να γίνει μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση, ένα χρόνος είναι λίγο. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω ένα μέσο όρο. Τουλάχιστον δύο έτη να είναι αυτή η παράταση, για να μπορέσουμε σε δύο χρόνια να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει επιστημονικός και με αποδεδειγμένο τρόπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά αφού άκουσα τα επιχειρήματα και τα θεμητά, τις θεμητές ε, παρατηρήσεις της ε, Ισπανίδας συναδέλφου θέλω να υπογραμμίσω τα εξή. γιατί και δικαίως είπε θα ήθελα να ε, μπορέσω να έχω μια τεκμηρίωση γιατί ο καθένας από εμά έχει να κάνει με τους ανθρώπους της περιφέρειάς του Δυστυχώς η συνάδελφος δεν άκουσε την αιτιολόγηση που έδωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής στην παρουσίασή της. Ήταν πληρέστατη από όλες τις πλευρές και εξήγησε ότι τα μέτρα που έλαβε η Ιταλική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια επέτρεψαν την μείωση κατά πολλές εκατοντάδες κιλά για κάθε αλίευμα και για κάθε σκάφος, πράγμα το οποίο επέφερε τα αποτελέσματα που στον κόλπο του Κάντιθ ε, επιτεύθηκαν μετά από το ε, ε, τα μέτρα που ελήφθησαν εκεί. Η Ιταλική κυβέρνηση λοιπόν στο αίτημά της για μείωση του μεγέθους διαπίστωσε και βρήκε λύσεις όπου στον κόλπο του Κάντιθ δυστυχώς ελήφθησαν καθυστερημένα γιατί όπως είπε η συνάδελφος υπήρχαν δυσκολίες γιατί οδηγούσαν ε, τα μέτρα που είχαν ληφθεί μέχρι τώρα σε μείωση του αποθέματος, δεν θα πρέπει να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Είμαστε σε, ένα, σε μια ενιαία αγορά. Δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε εμπορικού ε, τσακωμούς. Αλλά η τεχνική και επιστημονική δυνατότητα που διευκρινίστηκε από την Κομισιόν και που ε, μας ε, παρουσιάστηκε εδώ ενδελεχώς δεν οδηγεί σε καμία κανενός είδους λαβή για εμπορικό ε, πόλεμο. Η δική μας Επιτροπή είναι αρμόδια για την προστασία της αλληλείας. Δεν παρεσβρεί στην αξιολόγηση του ποια μπορεί να είναι, ποιος μπορεί να είναι ο ανταγωνισμός. Άρα λοιπόν εμείς οφείλουμε να αξιολογήσουμε μόνο εάν το απόθεμα κινδυνεύει από αυτού του είδους τη δραστηριότητα ή από την άλλη δραστηριότητα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πέρα από τα θεμητά συμφέροντα των ε, διαφόρων μας περιφερειών βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ε, που η Κομισιόν αντικειμενικά έδωσε ένα πλαίσιο για την πρόταση αυτή που έγινε. Και εγώ, όπως ο συνάδελφος Μιλάτζο και η συνάδελφος Κόντε, θεωρώ πως λόγω ακριβώς των επιστημονικών δεδομένων το ένα έτος μπορεί να παραταθεί σε δύο έτη για την εξαίρεση αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Mrs. Lenny, can you bring calm and reassurance? Κυρία Λένε, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε και να ηρεμήσετε την κατάσταση. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, προσπαθώ να κρατήσω την ηρεμία μου κι εγώ. ερχόμαι euh, ε, συχνά σε επαφή με την κυρία Γιγέρα. Την ευχαριστώ για το πάθος της για την αλληλεία και το οποίο και εγώ ε, μοιράζομαι μαζί της. Όπως σας είπα εδώ, πρόκειται απλά για εφαρμογή του βασικού κανονισμού, ο οποίος, ε, όπως και ο κανονισμός για τα τεχνικά μέτρα για τη Μεσόγειο, προβλέπει ότι στην περίπτωση ενός σχεδίου απόρριψης είναι δυνατόν να έχουμε εξαίρεση από το ελάχιστο μέγεθος, εάν αυτή η εξαίρεση δεν επηρεάζει το στόχο της βιώσιμης λίευση, δηλαδή της βιωσιμότητα του αποθέματος. Εάν υπάρχει πρόβλημα για την βιωσιμότητα του αποθέματος, δεν μπορούμε να μειώσουμε το, κι άλλο το μελάχιστο μέγεθο. Ε, λοιπόν είπαμε και στον Ιταλό Υπουργό και στον Ισπανό Υπουργό ότι η Κομισιόν θα, θα ακολουθούσε την, άποψη του επιστημονικού... της επιστημονικής ομάδας. Η Ιταλική κυβέρνηση και οι Ιταλικοί φορείς ε, κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να πλαισιώσουν αυτό το απόθεμα. Ε, όπως σας είπα, έφτιαξαν ένα σύστημα ελέγχου ε, και θαλάσσιο. Έχουν ξεπεράσει τους κανόνες του κανονισμού περί ελέγχων. Έχουν ε, φτιάξει ένα, τη δυνατότητα να, να παράγεται το στόκ σε καλές συνθήκες, έχουν φτιάξει σύστημα πιστοποίησης, μείωσαν τι ε, αλλιεύματα, ε, περιόρισαν δηλαδή ε, τις δυνατότητες αλλιεύματος και πρέπει να διαπιστώσουμε ότι λήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα, ότι οι φορείς πραγματικά υλοποιούν αυτά τα μέτρα Μάλιστα η Κομισιόν έκανε επιθεώρηση για να πάει να επαληθεύσει ότι όλες οι δεσμεύσεις τη ιταλική κυβέρνηση σε σχέση με τη διαχείριση αυτού του αποθέματος είχαν τηρηθεί και όντω έτσι συμβαίνει. Είχαμε όρους που είχε απαριθμίσει η Ιταλική κυβέρνηση για τα τεχνικά μέτρα, για τα μέτρα επιλεξιμότητας, για τα μέτρα ελέγχου, τα μέτρα διαχείρισης του στόκ και, ε, τα, και επιπρόσθετα μέτρα και ε, τα επαληθεύσαμε όλα και διαπιστώσαμε πως είχαν εφαρμοστεί επιτόπου. Επίσης διαπιστώσαμε πως η Ιταλία είχε φτιάξει ένα καθεστώς και μέτρα ερευνητικά για να βελτιώσει την επιλεξιμότητα των σειρώμενων ε, δικτυών και βλέπουμε ποιες προσπάθειες λοιπόν έκαναν οι φορείς για να βελτιώσουν την μηχανική διαλογή σε αυτό το είδος ότι ρίχνονται και πάλι στο νερό οι μικρότερες αχιβάδες ώστε ε, να μην επηρεάζεται η ο κύκλος της ζωής τους. Διαπιστώσαμε ποιες προσπάθειες λοιπόν έχουν γίνει ώστε αυτό το στόκ να αλλιεύεται με βιώσιμο τρόπο και ακριβώς η εξαίρεση στο ελάχιστο μέγεθος ε, διαπιστώσαμε πως το ελάχιστο μέγεθος που ζητείται μέσω αυτής της εξαίρεσης είναι, είναι πάνω από το μέγεθος ε, που, ε, στο οποίο γίνεται η αναπαραγωγή, που είναι 11 με 12 χιλιοστά, ενώ εδώ ζητείται το όριο των 22 χιλιοστών. Σε συμφωνία με την Ιταλική κυβέρνηση, λοιπόν, ε, είπαμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη περισσότερες μελέτες και βελτίωση της επιλεξιμότητας ε, στην διαλογή και ε, η πρόταση για τον ένα χρόνο προέρχεται από την Ιταλική κυβέρνηση την ίδια, γιατί η Ιταλική κυβέρνηση δέχτηκε η κατεξοδότηση αυτή πράξη να έχει διάρκεια ζωής μόνο ενός έτους, ώστε μετά να εφαρμοστεί ο κανονισμός με τα τεχνικά μέτρα. Στο μέλλον, αυτός ο κανονισμός που υιοθετήθηκε 14 Αυγούστου 2019, προβλέπει τη δυνατότητα στο μέλλον υιοθέτησης εξαίρεσης για τα ελάχιστα μεγέθη και γι' αυτό το λόγο έτσι ώστε ακόμα μια φορά να μπορέσουν να βελτιωθούν οι μελέτες επιστημονικές για αυτό το αποθεματικό και να μπορέσουν τον επόμενο χρόνο, αν το επιθυμεί η Ιταλική κυβέρνηση, να προτείνει μια νέα εξαίρεση μέσα στο κανονικό πλαίσιο του κανονισμού ε, των τεχνικών μέτρων, προτείνουμε για ένα έτος αυτή την ε, ε, εξαίρεση. Σε συμφωνία λοιπόν με τον Επίτροπο και την Ιταλική Κυβέρνηση πιστεύω πως είναι η καλύτερη προσέγγιση γιατί αυτό θα επιτρέψει την ενίσχυση της έρευνας, την ενίσχυση της επιλεξιμότητας, να δούμε ποιες είναι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα και έπειτα του χρόνου μέσα στο κανονικό πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού τεχνικών μέτρων να γίνει η αξιολόγηση αυτής της πιθανής εξαίρεσης για αυτό το είδος. Αυτά κύριε Πρόεδρε, κατανοώ τις παρατηρήσεις της κυρίας Αγγιλέρα, αλλά εδώ η Κομισιόν δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να εφαρμόσει τον κανονισμό για τη Μεσόγειο και το βασικό κανονισμό. Δεν ξέρω αν αυτό κάπως θα ε, ε, σας ηρεμήσει, αλλά πάντως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν είναι σύμφωνη με αυτά που παρουσίασε και στην Ιταλική και στην Ισπανική κυβέρνηση, δηλαδή να λάβει μια απόφαση επί τη βάση των επιστημονικών μελετών και των προσπαθειών που έκανε η Ιταλική κυβέρνηση για να πλαισιώσει αυτό τον στόλο. This is going to be ε, θα είστε σύντομοι, ελπίζω. Μάλιστα, Πρόεδρε. Λυπούμε λοιπόν, που παρατείνω αυτή τη διαδικασία λήψη απόφαση. Έχουμε χρόνο, δεν είναι ανάγκη να πάρουμε σήμερα την απόφαση, αλλά θα ήθελα να ζητήσω μια διευκρινήση, επειδή ε, αναφέρεστε σε μια κοινή δήλωση. Σύμφωνα με τη διαδικασία. Όμως εδώ είναι μόνο το αίτημα της Ιταλικής ε, κυβέρνησης. Άρα δεν είναι κοινή δήλωση. Δεν ξέρω. Ε. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιες διευκρινήσεις για αυτό το θέμα, να ξέρω αν ήθιστε αυτό ή όχι. Δεν ξέρω αν τεχνικά είναι σωστό ή όχι. Για να είμαι δίκαιος πρέπει να πω, είπε ότι και η Ισπανική κυβέρνηση και η Ιταλική κυβέρνηση ε, συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε. Ναι σε, σχέση με αυτή την υπόθεση της ε, κατεξοδότηση πράξη βασίζεται σε σύσταση που σύστησε η Ιταλική κυβέρνηση γιατί αφορά μόνο τα Ιταλικά χωρικά ύδατα. Αυτά τα ελάχιστα μεγέθη και υποχρέωση διατήρησης δεν αφορά παρά μόνο τα Ιταλικά χωρικά ύδατα. Ε, ήδη την πρώτη φορά όταν υιοθετήσαμε αυτή την ε, κατοξιδότηση πράξη, για την δεύτερη φορά που σας το προτείνουμε, επαληθεύσαμε με την νομική μας υπηρεσία αν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο και όντως όταν υπάρχει ένα απόθεμα το οποίο αφορά μόνο ένα ε, κράτος, μόνο έναν συγκεκριμένο στόλο που αλλιεύει στα συγκεκριμένα ύδατα, μια χώρα μπορεί να κάνει μια κοινή σύσταση για να ζητήσει σχέδιο απόρριψης για τα δικά του χωρικά ύδατα. Αυτή είναι η νομική ανάλυση που έγινε την προεπισμένη φορά και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και γι' αυτό το λόγο εδώ αυτή η κοινή δήλωση γίνεται μόνο από την Ιταλική κυβέρνηση για τα Ιταλικά χωρικά είδατα και για το συγκεκριμένο στόλο αποκλειστικά. Σας ευχαριστώ. Ήταν καλή αυτή η διευκρινήση. Κυρία Αγγιλέρα, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, δεν θέλετε. Εντάξει, αν θέλετε κάτι να καταθέσετε βεβαίως μπορείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ε, έχουμε και τον κανονισμό περί ICAT. Ε, δεν νομίζω να είναι επίμαχο το θέμα. Υπάρχει κάποιος που θέλει να μιλήσει. Κύριε Μαλίδα, θέλετε τον λόγο. Α, εντάξει, μάλιστα, ωραία. Έχετε λοιπόν τον λόγο. Σύντομη, σύντομη παρουσίαση παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσω για τον κανονισμό αυτόν που εγκρίθηκε στις 10 Ιουλίου. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, ο κανονισμός αυτός ε, τροποποιεί έναν υφιστάμενο κανονισμό, μια υφιστάμενη πολιτική. Ο βασικός ε, στόχος είναι να ενσωματωθούν ε, κάποιες συστάσεις τη σύστασης 1802 ε, που αφορούν ε, τον Ερυθρό μια επιτυχία της ε, ΑΕΚΑΤ στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε έναν ρόλο κλειδί, εάν μου επιτρέπετε. Ο κανονισμός αυτός βασίζεται σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους και επιβλήθη μετά από δικό τους αίτημα. Έχει σημαντικές ε, βελτιώσεις, ε, μειώνει τον αριθμό απορρίψεων, εγγυάται και την κερδοφορία των μικρών ψαράδων, εγγυάται ίσους όρους ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα άλλα συμβαλόμενα μέρη Τελειώνω λοιπόν. Δεν θα μπω στις τεχνικές λεπτομέρειες. Και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω να βλέπω κάποιον να θέλει να κάνει ερωτήσεις. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. στο σημείο 12, ανακοινώσεις ε, του Προέδρου για τις συστάσεις των συντονιστών από την πρωινή συνεδρίαση. Τις έχετε λάβει με email, αν έχετε ερωτήσεις, αντιρρήσεις. Εδώ πέρα ο Κλαούντιο κάνει ό,τι θέλει και αποφασίζει ουσιαστικά. Ε, πάντα έτσι ήταν. Μόνο οι συντονιστέ μόνο μόνο. Αν δεν υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις εγκρίνονται. Συστάσεις 13 ε, διάφορα δεν έχουμε κάτι. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου το απόγευμα και την επόμενη μέρα, πρωί και απόγευμα. Ο πρώτο ευχαριστή τους Ιερμηνείς, ευχαριστούμε και εμείς. Λύεται η συνεδρίαση.